Allora, buonasera a tutti, se prendete posto per favore. Allora, innanzitutto... Λοιπόν, πάνω απ' όλα, Κάνω μια αλλαγή όσον αφορά την έγκριση του σχεδίου μερίσια διάταξη. Μετά την παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεω του κυρίου Λιμπεράτσκι, η Επιτροπή Άνκετ Άντορ θα παρουσιάσω στη συνεδρίαση μια έκθεση για τις αρχικές συνέπειες του σχεδίου δράσης για την εποπτεία, για την εφαρμογή της εποπτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κοινή διαχείριση των θετικών ε, δράσεων. Θα αλλάξει το σημείο 5 τη ημερήσιας διάταξη. Έχουμε τους αν και άντο του επιτρόπους εδώ. Και η συζήτηση θα διαρκέσει μία ώρα. Όσον αφορά το σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης, τα πρακτικά 2 και 3 Δεκεμβρίου του 2009, τα πρακτικά τη συνεδρίασης 25, 26, 27, 28 Ιανουαρίου, όλα αυτά θα σας προσταλούμε στο ηλεκτρονικού ταχυδρομείο. Ξέρετε τις γλώσσε, μεταδίδεται μέσω web streaming τη συνεδρίαση. Αύριο το πρωί φέρτε τις κάρτες ψηφοφορίες για ψηφοφορία. Όσον αφορά τη διαδικασία που έχουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Χαιρετίζουμε τον Υπουργό Οικονομικά. Καλώς σου Πανιά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εφόσον θα μιλήσει πρώτα ο κύριος Υπουργός, Ισπανός Υπουργός, θα έλεγα ξεκινήσουμε τον ακούσουμε για να μην χρονοτριβούμε, θα φτάσει και ο κύριος Λιμπεράκης και εντωμεταξύ και θα του δώσουμε το λόγο όσον αφορά τι απαλλαγέ του 2008 και τι συστάσει του Συμβουλίου, δίνω το λόγο στον Υπουργό Κάρλο Ογκάνια, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ για να εκπροσωπώ το Συμβούλιο και να σας παρουσιάσω τις συστάσεις για την έγκριση της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προπολογισμό του 2008. Μετά από την έγκριση του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ απεστάλησαν τα έγγραφα στις 16 Φεβρουαρίου. Τους τελευταίους μήνες το Συμβούλιο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 Λοιπόν, όσον αφορά την έκθεση του 2008, λοιπόν, αναγνωρίστηκε ε, από πλευρά ε, του Λεκτικού Συνεδρίου ότι έγινε βελτίωση στη διαχείριση των πόρων Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορου τομεί πολιτική, κυρίω για τη γεωργία και για του ε, φυσικού πόρου. Όμω, θα πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές και να καταλάβουμε ότι οι προσπάθειες που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κάτι μέλη προς βελτίωση της εχειρήσεως των πόρων δεν δείχνουν άμεσα αποτελέσματα πάντα και παρατηρητέα αποτελέσματα. Σε εκπληστεί ότι η δήλωση το δελτίο αξιοπιστίας παρέμεινε αρνητικό για ένα σημαντικό τμήμα του προπολογισμού και το 2008 Λοιπόν, για ποιο λόγο έκαναν τις συστάσεις που έκαναν στο Συμβούλιο για την χορήγηση τη απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να αναφέρω του ετήσιου λογαριασμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, όπου εκεί σημειώνεται με ικανοποίηση ότι για δεύτερη χρονιά το ελεκτικό συνέδριο ε, τοποθετήθηκε θετικά όσον αφορά την εξοπιστία των στοιχείων και παραδέχτηκε ότι παρουσιάζουν σωστά την οικονομική θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αναγνωρίζει το Συμβούλιο την ε, σωστή παρουσίαση των στοιχείων και τη ομαδοποίησης των λογιστικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν ε, και ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρατήσει αυτό το επίπεδο των στοιχείων της, ε, των λογιστικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το κατά πόσο έγιναν σωστά οι συναλλαγές και κατά πόσο λειτουργήσαν σωστά τα συστήματα τα υποπτικά. Το Συμβούλιο είναι ικανοποιημένο ε, με την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου για τα εισοδήματα και την ανάληψη υποχρεώσεων σε όλους τους τομείς και για τις πληρωμές στον τομέα της παιδείας, ε, ε, και διοίκηση γενικά και το Συμβούλιο καλωσορίζει τις ορατές βελτιώσεις που έγιναν στο γεωργικό τομέα και στον τομέα των φυσικών πόρων για τις πληρωμές σε αυτόν τον τομέα έγινε μια, μια εκτίμηση σφάλματος που ήταν κάτω από το αντικειμενικό κριτήριο το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διοίκησης που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών όσον αφορά το τομέα εγγυήσεων από του ΦΕΟΚΑ θεωρείται ότι βελτιώθηκε ο τομέας αυτό. Σημαντικό βήμα είναι αυτό, λέει το Συμβούλιο, για την καλύτερη οικονομική διαχείριση. Μόνο λόγω των μεγαλύτερων επιπέδων σφαλμάτων που διαπιστώνονται στον τομέα δαπανών για την ε, βελτίωση της υπαίθρου, εκεί ε, έδωσε, έθεσε κάποιους όρους όσον αφορά την γνωμοδότηση του το ελεγκτικό συνέδριο, διαπιστώντα ταυτόχρονα κάποιε προόδου. Παρά τα θετικά μηνύματα, εξακολούθησε να επηρεάζεται από σφάλματα το τομέα των δαπανών. Σε σημαντικούς τομείς πολιτικής εντοπίστηκαν μόνο ορισμένες μειωμένες βελτιώσεις και το ελεκτικό συνέδριο έχει αρνητική άποψη όσον αφορά την έρευνα, ενέργεια, συνοχή, μεταφορές, εξωτερική ανάπτυξη, εξωτερικής βοήθειας, ανάπτυξη και διεύρυνση και εκφράζει τη λύπη του γι' αυτό και ενθαρρύνει όλους τους φορείς να καταβάλουν ε, προσπάθειες σχετικά με αυτό και θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτούς τους τομείς, να μειωθούν οι ατασταλίες και τα προβλήματα και τα αποτελέσματα να είναι πιο αποδεκτά, να είναι καλύτερα. Το Συμβούλιο ανησυχεί όλο ιδιαίτερο για την εκτίμηση του ελεκτικού συνεδρίου ότι στον τομέα τη συνοχή το 11% των συνολικών ποσών δεν θα έπρεπε να επιστραφεί. Όμως να προσθέσω ότι αυτό το στοιχείο αφορά επιστροφές σε προγράμματα πολιτικής συνοχής της προτέρα προγραμματικής περίοδου 2000 με 2006 που όπως γνωρίζουμε επηρεάστηκε πολύ από συστημικά σφάλματα. Οι βελτιωμένες δομές εποπτείες όσον αφορά τους κανονισμούς για την νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 μπορεί να αξιολογηθεί μόνο όταν οι επιστροφές από αυτά τα προγράμματα θα αρχίσουν να θα αποτελέσουν δικείμενο ελέγχων. Επιπλέον, ο πολιτής χαρακτήρας των δαπανών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι ατασταλίες που ενετόπισε το ε, ελεκτικό συνέδριο είναι προβλήματα επιλεξιμότητας που μέσω ανακτήσεων και διορθώσεων μπορούν να καλυφθούν αυτά τα σφάλματα τα επόμενα χρόνια. Ε, σε μεγάλο ποσοστό όλα αυτά έχουν γίνει προσπάθειες, διότι μιλάμε για το 2008 και το Συμβούλιο σημειώνει το ελεκτικό συνέδριο δεν ανέφερε καμία περίπτωση ενδεχομένης απάτης. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αντιδράσουν κατεπηγόντως από τη στιγμή που θα φανούν τα προβλήματα. Να βελτιωθεί η εποπτεία, οι διαγωνισμοί, ο έλεγχος της εκτέλεσης και να γίνουν κάποιες ορθωτικές κινήσεις. Επίσης, το Συμβούλιο αυτό. Λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια αξιόπιστη μηχανισμοί και αποτελεσματική, γιατί αυτό πάνε να πει αποτελεσματικό έλεγχο. Άρα θα πρέπει προ όλε αυτέ τι κατευθύνσει να έχουμε μία καλύτερη εφαρμογή, απλούστευση των ε, κανόνων που σήμερα διέπονται από την πολυνομία, την περιπλοκότητα και μόλι έχουμε επομένω αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι θα πρέπει οι διατάξεις να είναι κατανοητές, ξεκάθαρες και να είναι ομοιογενείς η εφαρμογή τους. Απλούστευση να γίνει όσον αφορά την σημερινή για τον προγραμματισμό να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες όταν ήρθε η ώρα εκπόνησης των προγραμμάτων για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε σχέση με αυτό επίσης υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ αυτών των διατάξεων αλλά και των προβλέψεων των δαπανών τόσο ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Εξάλλου χρειάζεται αρκετός έλεγχος ούτως ώστε να υπάρχουν εγγύσεις για μια χρηστή υγιή διαχείριση των πόρων. Είμαι θα πεπισμένοι ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και αποτελεσματική σε αυτούς τους ελέγχους. Επίσης θα πρέπει να, είναι, να υπάρχει αναλογία μεταξύ ένταση ελέγχων και αποτελεσμάτων αυτών. Και θα πρέπει επίση τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν περισσότερο τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και να υπάρχει ανταλλαγή των υπαρχουσών πληροφοριών στο βαθμό του δυνατού. Επίση, θα πρέπει να έχουμε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τον οικονομικό έλεγχο σε κάθε επίπεδο. Και έτσι να μην έχουμε επικαλύψεις έτσι να υπάρχει μια κοινή αντίληψη για τους εν λόγω οικονομικούς ελέγχους τώρα. Οι βελτιώσεις όσον αφορά τα ταμεία, όπως έχει πει και το ελεκτικό συνέδριο, υπόσχονται πολλά όσον αφορά το ότι θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να κάνουμε βήματα πρόοδου. Όμω, για να μπορέσουμε αυτό το στόχο να τον πετύχουμε, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι η Κομισιόν δηλαδή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να βοηθήσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να πετύχουμε το βασικό μας στόχο. Θετικό δάση. Είναι κατακλείδη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων της Ένωσης. Όμως, αν λάβουμε υπόψη όλες τις μεταβλητές θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα της χρήσης του 2008. Εν τέλει, θα σας πω ότι έχουμε το θέμα της έγκρισης των 23 οργανισμών και υπηρεσιών των νομικών προσώπων της Νομικής Ένωσης. Έτσι θεωρούμε ότι υπάρχει συμβολή στη διαχείριση του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι συνιστά το Ελληνικό Συνέδριο τόσο ώστε να βελτιωθεί αυτή η διαχείριση. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιωθεί η διαχείριση των, ε, των, των κοινών ε, εγχειρημάτων, των, των υπηρεσιών, όπως πει το Ελληνικό Συνέδριο, για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση που έχει συστήσει, χωρίς καμία επιφύλαξη και δισταγμό. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λιμπεράτσκι, έχετε το λόγο.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 το ελεκτικό συνέδριο παρουσίασε σύνοψη. Παρουσίασε τις αλλαγές της καταστάσεως. Και μας είπε τι μεταβολές έχουν επέλθει όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Τι υπάρχει πρόβλημα, λέει και ο πρόεδρος, με, την, με, την, ε, με το αγγλικό κανάλι διερμηνίας. υπάρχει τεχνικό πρόβλημα εδώ. Λοιπόν, Πρέπει να πω ότι στην περίοδο που συζητάμε είδαμε βελτιώσεις όσον αφορά τα σφάλματα. 2% ε, ήταν τα σφάλματα. Διακόπτεται εδώ η Γερμανία και από άλλα κανάλια. Ah uh, Ξαναρχίζει. Κυρίες και κύριοι, τι έχουμε εδώ. 47 όσον αφορά τις δαπάνε. Οπότε, επαναλαμβάνω, 47% των δαπανών βρίσκεται κάτω από αυτό το 2% του ετησίου περιθωρίου και επομένως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση στην κατάσταση. 57% βρίσκεται πάνω από το όριο. Επομένως με αυτό το ρυθμό πάμε για μια 20 για την ακρίβεια 20 χρόνια και 3 μήνες ούτω ώστε ο προϋπολογισμός να βρίσκεται κάτω από το όριο αυτού του ετησίου 2%. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Επομένως, η ταχύτητα, ο ρυθμός πρόοδου είναι πολύ σημαντικός. Τώρα υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Πρόκειται για τα ποσά εκείνα τα οποία μεταφέρονται από τη μία χρονιά στην άλλη 30% ή 155 δις ευρώ. Εμείς δε, ως Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο μας οδηγεί σε ένα άλλο χρήσιμο συμπέρασμα. Δηλαδή, δεχόμενα έτσι, δεν μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα όσο μπορούμε από τον προπολογισμό της Ένωσης. Και σας τονίζω επομένω ότι έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά τα εγκάρσια ή οριζόντια ζητήματα. Και αυτό το οποίο απορρέει από την ε, ανάλυση που έκανα είναι μια θετική τάση. Η ανωδική 0,4%. Συν 0,4% όσον αφορά τη μείωση σε παιδεία, γεωργία, μεταφορές και άλλα. Εις δε το σημείο 5 διατυπώνουμε το ότι δυστυχώς ακόμα θα πρέπει να κάνουμε πολλά όσον αφορά τις ε, αντικανονικότητες, τις παρανομίες, τις παρατυπίες, όσον αφορά τα ταμεία, όσον αφορά τις εξωτερικέ δράσεις τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δουλεύει συλλογικά ως σώμα και να μην δρά από μόνος του κάθε επίτροπος. Άρα, σας υπενθυμίζω ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές επιφυλάξεις όσον αφορά τον προπολογισμό και τις διατυπώνουμε στην διάταξη 15 έως και 18. Επιφυλάξεις δε αυτές που σχετίζονται με διαφορά όσον αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων και τον τρόπο που καλύπτονται αφορούν αυτά τα ποσά τα οποία μεταφέρονται. Αυτά τα 155 δις και είναι επομένω κάτι το οποίο μας προβληματίζει σοβαρά. Τόσο αφορά την ανάκτηση, ιδίω όσον αφορά τα διαρθωτικά ταμεία, είναι θέμα που μας έχει απασχολήσει και προηγουμένως. Οπότε Βεβαίως ξέρουμε ότι το έργο εδώ που έχουμε λάβει είναι δύσκολο και ξέρουμε και από το παρελθόν ότι είναι περίπλοκες διαδικασίες. Πάντως, σας παραπέμπω στην διάταξη υπαριθμών 21, οπότε και να απευθύνουμε έγκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να υποβάλει ένα αποτελεσματικό σύστημα, σύστημα πολιετές, όσον αφορά την ανάκτηση των ποσών που θέλουμε και εκεί να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες του κάθε κράτου Επίσης, Θέλουμε πάρα πολύ θετικό το ότι η Επιτροπή δέχθηκε τις ντάσεις των κρατών μελών. Όμως, η καθεμιά είναι διαφορετική. Η καθεμιά ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία. Τα χρονικά πλαίσια είναι σαφή, ούτε επίσης το τι, ποια είναι τα ποσά αναφορά σε κάθε περίοδο αναφοράς. Άρα τα πράγματα εδώ είναι κάπως θολά και γι' αυτό λέμε ότι η Κομισιόν καλά έκανε και φρόντισε να υπάρχουν αυτές, όμως χρειάζεται να βρεθεί μια μεθοδολογία ενιαία. Θέλουμε όλα τα κρατημέλη να υποβάλουν τις ντάς δυνάμει κοινών διατάξεων και κανόνων. Τώρα, στον αφορά του εσωτερικού οικονομολόγου στην Κομισιόν, ήδη έχει γίνει μια σχετική συζήτηση και ε, συναντηθήκαμε 14 φορέ. Και με επιτρόπου και με γενικού διευθυντέ. Οπότε και συζητήσαμε για τα θέματα αυτού του στήματο οικονομικού ελέγχου τη Κομισιόν και βέβαια δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε για το ότι θα πρέπει να έχει κριτήριο την απόδοση το αποτέλεσμα η Κομισιόν δεν είναι δυνατόν να, μετατραπεί σε ένα δεύτερο ελληνικό συνέδριο. Όμως, όμως, Κάποιες γενικές διευθύνσεις θα πάνε καλύτερα. Κάποιες βελτιώθηκαν, αλλά κάποιες άλλες όμως έχουν κάνει πισωγύρισμα, επομένως έχουμε ακόμα διαφοροποιημένες επιδόσεις. Επίσης, απλώς κοινοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντικό στην έκθεση η πολιτική και διοικητική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Αλλά να λάβουμε και τους στόχους της Ένωσης και τελικά του και του Κοινοβουλίου. με τους οποίους στόχους θα πρέπει να είναι σύντονοι βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναφέρουμε πιο συγκεκριμένε εξωτερικέ δράσει αλλά και τα διάφορα ταμεία τη Ένωση. Επομένω, αυτέ οι επιφυλάξει μα διατυπώνονται σε περισσότερα σημεία. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Και ο Μιλών έχει αναλάβει να συντάξει αυτό το κείμενο και ως συμπέρασμα πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν μάλλον συμφωνεί με τις επιφυλάξεις μας. Όμως, βελτιώσεις δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε υπάρχει συνέχεια από πλευράς τους. Δεν έχουν πετύχει κανένα συγκεκριμένο στόχο που έχει μπει. Και γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε δύο σημεία που ακόμα δεν τα έχω εντάξει στο σώμα του κειμένου. Πρώτον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, έχουν επιφέρει κάποιες δηλώσεις ε, οι οποίες σιγά σιγά προχωρούν όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών. Οπότε η απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί. Δεύτερο συμπέρασμα. Λάβετε το και αυτό υπόψη. Θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάτσουμε και να φτιάξουμε ένα εργασία σε ένα πρόγραμμα δράσης, ούτω ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα οριζόντια θέματα. Τη διαχείριση του προπολογισμού, τις εθνικές δηλώσεις τον εσωτερικό οικονομικό έλεγχο της Κομισιόν, τα της πολιτικής και διοικητικής ευθύνης που φέρει η Κομισιόν, το πολιετές πρόγραμμα ανάκτησης και να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον μας στο Ταμείο Συνοχής αλλά και στις εξωτερικές δράσεις. Όταν δεν καταλήξει κάποιο χρονικό πλαίσιο η Κομισιόν όσον αφορά το πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να εκπονήσουμε αυτό το πρόγραμμα δράσης, και όταν μας το υποβάλλει τότε να επανέλθουμε στην συζήτηση της απαλλαγής. Θα τη δώσουμε δηλαδή ή δεν τη δώσουμε. Παρακαλώ τώρα να τα σκεφτούν όλα αυτά οι συνάδελφοι διότι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια τοποθέτηση. Και θα ήθελα ταχαίως να δω αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοποίηση των ενωσιακών πόρων. Να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Όσον αφορά το πού πάνε τα χρήματα. Να έχουμε value for money, να πιάνουν τόπο. Και θέλουμε πάρα πολύ εντυπωσιακέ βελτιώσει όσον αφορά τη μεσονομική πειθαρχία και τι δαπάνε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν καθυστερήσεις που είναι σημαντικές όσον αφορά τις πιστός πληρωμών να σταματήσουν. Αυτό είναι υπόσχεση, δέσμευση όλων των κρατών μελών. Και αν δεν μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, τότε απονευρώνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί πιο αποτελεσματικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το καλό όλων. Σας ευχαριστώ κύριε Λιμπεράλσκι. Να δώσω το λόγο στους βουλευτές. Το Συμβούλιο θέλει να ακούσει πρώτα μια ομάδα απαντήσεων και να απαντήσει μετά ομαδικά. Στάις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που ο κύριος Λιμπεράτσκι εξήγησε με σαφήνεια και ακρίβεια το πώς θα προχωρήσει για το θέμα της απαλλαγής της Κομισιόν. Και μάλιστα παρουσία και του κυρίου Υφυπουργού. Βρίσκω ότι είναι σωστό διότι η σοβαρότητα με την οποία εγκύπτουν Κοινοβούλιο και Επιτροπή σε αυτή την υπόθεση απαλλαγής της Επιτροπής είναι σημαντική. Εδώ και δέκα χρόνια που είμαι Ευρωβουλευτής έχω την εντύπωση μέχρι τώρα και είναι η δεύτερη απαλλαγή στην οποία ε, συμμετέχω έχω την εντύπωση ότι το Συμβούλιο των Υπουργών δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα σοβαρά. Βλέποντας την, εξετάζοντας την έκθεση του ελεγκτικού Συμβουλίου διαπιστώνει κανείς ότι λέει ότι 31% του προϋπολογισμού εκτελείται με ένα περιθώριο σφάλματος τουλάχιστον 5%. Αυτό σημαίνει ότι το περιθώριο σφάλματος συνήθως είναι παραπάνω. Και αν τώρα εξετάσουμε τα διάφορα διορθωτικά ταμεία, βλέπουμε να αναφέρεται και περιθώριο σφάλματος 11%. Εδώ και χρόνια, όχι μόνο η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού έχει την πεποίθηση αλλά και ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα ε, το συζητήσαμε και στην Ολομέλεια ότι είναι μοιρασμένε οι ευθύνε με την έννοια ότι μεγάλο μέρος του προπολογισμού εκτελείται κοινή ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών μελών. και είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση των χρημάτων. Ως Επιτροπή Ελέγχου του Προεπορισμού αλλά και ως ε, Κοινοβούλιο γενικότερα έχουμε κατά επανάληψη πει ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σύστημα όπου κάθε χώρα μέλος και εν τέλει βέβαια οι Υπουργοί Οικονομικών της κάθε χώρας μέλους να υποχρεούνται να πιστοποιούν ότι με τα μέσα που του διατέθηκαν, τα μέσα μάλλον που τα, δηλαδή τα κονδύλια που του διατέθηκαν, τα διαχειρίστηκε ορθώς, ε, εξέτασε τον τρόπο και ελέγξε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείρισή τους και ότι η διαχείριση αυτή ήταν ορθή για τον λόγο αυτό, ο λόγο υπουργό πιστοποιεί ότι έγινε σωστή διαχείριση. Βέβαια, η πρότασή μα αυτή δεν έχει τύχη τη εγκρίσεω του Συμβουλίου. Λίγε χώρε μέλη, ίσω οι χώρε των λεγόμενων ευρωσκεπτικιστών, είναι εκείνε που λένε ότι α, ναι, το δοκιμάσουμε. Άκουσα, κύριε Υπουργέ, ότι και ο Βέλγος Υπουργός ο Βέργος Υπουργός είναι κατά της απαλλαγής. Ή μάλλον ο Ολλανδός Υπουργός. Θα ήθελα να μάθω αν αυτό αληθεύει. Επίσης, υποτίθεται ότι θα διεξαχθεί αυτή η συζήτηση στο Συμβούλιο υποτίθεται ότι υπάρχουν, έχουν διαπιστωθεί κάποιες ανομαλίες, ότι έχουν γίνει πολλά σφάλματα, έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις ή γίνονται σχετικές δηλώσεις, αλλά τα πράγματα παραμένουν στα ίδια. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω εάν εσείς ως αρμόδιος υπουργό θα φροντίσετε να υλοποιηθούν αυτά που ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί στη συνεργασία με τους... Κοιτάξτε, Κρατούν πολλοί ερωτήσεις, έχουμε πολλά ακόμα θέματα, έχουμε πέντε ερωτήσεις, δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Παρακαλώ πάρα πολύ να μην είστε τόσο λύση. Κυρία Γκρέσ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, διαβάζοντας, διαβάζοντας το ε, κείμενο της έκθεσης του Συμβουλίου έχει κανείς την εντύπωση ότι ε, πρόκειται για ένα είδος σάτυρας διότι τα προβλήματα διαπιστώνονται στην εκτέλεση του προπολογισμού στι χώρε μέλη και το Συμβούλιο παριστάνει εδώ σαν δήθεν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, τι πρόκειται να κάνει το Συμβούλιο για να μπορέσει να βελτιωθεί η διαχείριση και να βελτιωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς άλλωστε εκπροσωπείτε μια ενδιαφέρουσα χώρα μέλος η οποία έχει ενδιαφέρον από την, από την άποψη ότι 60% των κακών ε, διαχειρήσεων των σφαλμάτων δηλαδή εντοπίζονται στην Ισπανία και 95% συνολικά Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποιον μεμφόμαστε. Από την Ισπανία θα πρέπει να ακούσουμε λοιπόν ξεκάθαρα λόγια. Ποια διδάγματα αντλείτε εσείς. Για παράδειγμα, ε, έχετε δεχθεί ότι η οδηγία για τους δημόσιους διαγωνισμούς, δημόσιες προμήθειες δηλαδή, έχει εφαρμοστεί εσφαλμένα στη χώρα σας ποια συμπεράσματα βγάζετε. Επίσης η Ισπανία δεν έχει συμμετάσχει στον διάλογο που έχουμε διεξαγάγει μέχρι τώρα εδώ για να μειωθούν τα ποσοστά σφαλμάτων. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι θα πράξει το Συμβούλιο Υπουργών για να βελτιωθεί η διαχείριση και τι θα πράξει ειδικότερα η Ισπανία. Ε, ευχαριστώ. Ο κ. Οντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κύριε Υπουργέ, όπως και συνάδελφοι, να πω ότι δεν αφορά το βασίλειο της Ισπανίας όλους ιδιαίτερα στο θέμα, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι το Συμβούλιο δεν, ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρεται επαρκώς όσον αφορά τις ανάγκες βελτιώσεως της διαχειρίσεως των ε, κοινοτικών πόρων και γνωρίζετε ότι 80% του προπολογισμού που είναι στην, είναι στην κοινή διαχείριση και θα θέλαμε σε αυτή την απαλλαγή για μία φορά το Συμβούλιο να δείξει βούληση, να είναι στο πλευρό μας ούτως ώστε ως αρχή του προϋπολογισμού να βελτιωθεί να συνεισφέρει να βοηθηθεί κατάσταση. Δεν έρχεστε ποτέ στην, δεν έρχεται στην Ολομέλεια όταν ήρθε το ελεκτικό συνέδριο να παρουσιάσει την εκθεσή του, θα έρθετε για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Θα ήταν ενδιαφέρον να δείξετε το ενδιαφέρον που έχετε. Λοιπόν, θέλουμε να τα ακούσουμε αυτό. Δεν ακούμε αυτή την αποφασιστικότητα σε αυτά που μα λέτε. Γιατί δεν βλέπουμε στα ψηφίσματά σα. Εκτιμώ το την εισηγητή, είναι πολύ την εισηγήτρια. Λοιπόν, όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς, έχουμε θετική τοποθέτηση του λεκτικού συνεδρίου, αλλά δεν υπάρχει σύσταση. Θεωρώ ότι η πολιτική συζήτηση περιμένει τοποθέτηση του εισηγητή. Δεν θα διευκολυνθεί η πολιτική συζήτηση, αλλά θα πρέπει να γίνει. Ερώτημα. Πώς βλέπετε, όπως είπε η κυρία Γκράσλε, το θέμα των εθνικών δηλώσεων. Ναι, ιού, κάποια μέρα θα τις έχουμε τις δηλώσεις και αν δεν τις έχουμε, τι προτείνει το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο μας έκανε προτάσεις για την απαλλαγή του περσινού έτους, κάναμε προτάσεις. Τι προτείνετε εσείς σε αντικατάσταση, αν δεν θέλετε, τις εθνικές δηλώσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Μπράντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου που μίλησαν πριν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε, να ζητούμε αυτές τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας που είναι σημαντικό ε, εργαλείο για να επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις χώρες μέλη. Προ λίγων εβδομάδων συμμετείχαμε στην Χάγη σε διάσκεψη με τα Εθνικά Κοινοβούλια και εκεί εκφράστηκε η επιθυμία για μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από τον κύριο Υπουργό πώς προτίθεται να το εφαρμόσει αυτό. Οι συνάδελφοί μου μίλησαν ήδη για τα θέματα αυτά. Εγώ θα πω πολύ σύντομα ότι άκουσα ότι στο Συμβούλιο ότι σχετικά με την δαπάνηση χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων στις χώρες μέλη ισχύει η αρχή της μη παρέμβασης. Δηλαδή δεν θίγονται τα κακοσκήμενα κατά κάποιο τρόπο. Εγώ το βρίσκω αυτό ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο διότι εάν γίνονταν συζητήσεις θα μπορούσαν να προκύψουν και βελτιώσεις. Φαίνεται σαν να μην ενδιαφέρονται καθόλου οι χώρες μέλη για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα άλλες χώρες μέλη. Αυτό δείχνει πραγματική αδιαφορία από πλευρά των χωρών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Υφυπουργό εάν η δαπάνηση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων στις χώρες μέλη δεν θα έπρεπε να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και να λάβει το λόγο κάθε χώρα μέλο και να προβεί σε δήλωση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα χρήματα. Άρα τότε θα μπορούσαν οι υπόλοιπε χώρες να ελέγξουν πολύ καλύτερα και να βελτιωθεί και η πειθαρχία περί τις δαπάνες αυτέ. Και ίσως τότε να καταλήγαμε κάποτε και στις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Οι κάτω χώρε δεν κατεψήφισαν την απαλλαγή, απέσχουν Αυτό διορθώνω για πριν. Τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν διαφορετικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που κατέβαλε για την έκθεση αυτή, για τη σύνταξή της. Όμως έχω αρκετές παρατηρήσεις που αφορούν τα θέματα, τα στομή για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Άρθρα 147 Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε όσον αφορά τα άρθρα. Να σε πιστήσω στην προσοχή σε κάτι, ότι πολλά σημαντικά βήματα ελήφθησαν στις χώρες μας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Πολλά σχέδια δράσης υιοθετήθηκαν και έγιναν διάφορες εκθέσεις συμμόρφωσης για τα λειτουργικά προγράμματα, πάγωσαν πολύ πόροι και παρακαλώ αυτό να το έχετε υπόψη στην τελική εκδοχή της εκθέσεώς σας διότι πιστεύω στην αντικειμενικότητα της Επιτροπής αυτής και του σώματος. Αν πρέπει να δούμε τα αρνητικά στοιχεία θα πρέπει να δεχτούμε και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Και ελπίζω αυτό να το έχετε υπόψη σας. Σας ευχαριστώ. Και ο Σγκέιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Υφυπουργέ, βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση εδώ ως ευρωβουλευτές. Είμαστε μέρος της αρχής του προϋπολογισμού, αλλά τα προβλήματα που διαπιστώνουμε στην διαχείριση, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού δεν μπορούμε πάντα να συζητήσουμε μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού βρίσκονται σε κοινή διαχείριση. Δηλαδή, συχνά στι συνομιλίε μας οι υπάλληλοι ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αξιωματούχοι τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε δεν τα διαχειριζόμαστε εμείς τα χρήματα αυτά. Εξετάζοντα τις δηλώσει σα ανακύπτει για μένα το ερώτημα πώ το Συμβούλιο, πώς κρίνει το Συμβούλιο τον αποφασιστικό ρόλο των χωρών μελών και πώς θα τον βελτιώσει. ενδιαφερόμαστε να προχωρήσουμε σε διάλογο, όχι μόνο τον διαρκή διάλογο που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με το Συμβούλιο, για να συζητήσουμε αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Ευρωπαϊκός προπολογισμό και στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή το υψηλό ποσοστό σφαλμάτων. Ο κύριος ε, Γκεμπράντι προηγουμένω είπε ότι και τα εθνικά κοινοβούλια ενδιαφέρονται, διότι εν τέλει στο κάτω της γραφής είναι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και τα χρήματα που έρχονται στη δική μου πατρίδα, τη Γερμανία, μπορεί να είναι χρήματα και από άλλους ε, φορολογούμενους, αλλά εν τέλει είναι και χρήματα Γερμανών φορολογουμένων και αυτοί ενδιαφέρονται. Δεν λέω ότι σέβομαι λιγότερο τα χρήματα των άλλων φορολογουμένων, των άλλων εθνών δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι τα βάζουν στο ίδιο καλάθι και από, όλα, και από αυτά αντλούμε. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε για παράδειγμα τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας, αξιοπιστίας ως ένα μέσον να εμφανίζονται τα πράγματα αυτά και ενώπιον του Συμβουλίου Υπουργών. Είναι η Ισπανική Προεδρία διατεθειμένη να προχωρήσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ζάντεργκεν. Ευχαριστώ πολύ. Ένα πολύ σύντομο ερώτημα, Υπουργέ. Σε συνάρτηση με αυτά που είπε ο κύριος Στάς, τι έγινε στη συνεδρία της Κορεπέρ, ελήφθη μια απόφαση από ό,τι καταλαβαίνω, να τεθεί τέρμα στην πρόταση για απαλλαγή. Υπήρξε χώρα που ήταν κατά, ψήφισε κατά, υπήρξε χώρη που απίσχε. Δεν είναι ανάγκη να κατονομάστε τη χώρα, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε να μας πει ο υπουργό αν υπήρχε κάποια χώρη που καταψήφισε ε, ή είχε απόσχει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Αγιάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, Υπουργό που ήρθε να συζητήσουμε και φυσικά έγινε συζήτηση στο Αντιποσυμβούλιο. Συμβούλιο για όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας, μας αφορούν γιατί αφορούν στην εκτέλεση του προπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γίνουν αυτές τις διορθώσεις όσον αφορά την πολιτική συνοχή, να μην μείνει καμία αμφιβολία, γιατί υπάρχουν σημαντικοί πόροι. Προέρχονται από την συγχρηματοδότηση, οπότε και το ένα κομμάτι και το άλλο της συγχρηματοδότησης θα πρέπει να διακρίνονται από διαφάνεια σε ένα τοπίο ξεκάθαρο. Λοιπόν, θα πρέπει να ενεργήσει αναλόγως η, Ισπανία που τώρα την Προεδρία και επομένω θα πρέπει να συνεχίσει με την ίδια επιτυχία την πολιτική της συνοχής όπως είχε γίνει και προηγουμένως από άλλους. Άρα θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στη διαχείριση των των πόρων. Μήπως μπορεί να μας πει το Συμβούλιο πώς μπορεί να βοηθήσει η Ισπανική Προεδρία για αυτό το στόχο. Το Βέλγιο, οι κάτω και το Βέλγιο κιόλας που έχει και ομοσπονδιακή δομή εν μέρη. Σε αυτές τις χώρες επομένως Τώρα υπάρχει προβληματισμός για το πώς θα υπάρχει περισσότερη αξιοποίηση των ε, πόρων, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερος έλεγχος. Και έτσι να δούμε για Γερμανία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, πώς μπορούμε να έχουμε κάποια βελτίωση. με κάποια αποκέντρωση να φτάνουν στον τελικό αποδέκτη τα χρήματα. Πεςτε μας, επί τη βάση της ζήτησης που έγινε στο άτυπο συμβούλιο, πώς μπορεί να βοηθήσει για όλα αυτά η Ισπανική Προεδρία. Γιατί πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν εξορθολογισμό της κατάστασης και της, ε, της ε, πολιτικής συνοχής. Πρόεδρος. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, να κάνω και εγώ ένα τελευταίο ερώτημα και μετά θα έχουμε ένα τέταρτο που για να απαντήσετε σε ερωτήσει. Πρόσφατα διαβάσαμε λοιπόν αυτό που έκανε το Νυχτικό Συνέδριο για τη χρήση 2008 και όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι πολλά είναι τα σφάλματα ακόμα, πολύ σοβαρά σφάλματα και πιστεύω σφάλματα που δείχνουν απάτες όπως το συζητήσαμε επανειλημμένα κυρίως όσον αφορά κάποια κάτι μέλη. Λοιπόν συγκεκριμένο ερώτημα, τι προτίθεται να κάνει το Συμβούλιο έναντι των κρατών μελών εκείνων που επί σειρά ετών τώρα και πολύ συχνά είναι υπεύθυνα για απάτες κατά της Ευρωπαϊκής σας Πώς προτίθεστε να ενισχύσετε την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων έναντι αυτών των κρατών μελών και πώς μπορείτε να εγγυηθείτε καλύτερα τη συνεργασία των ε, κρατών μελών αν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα χέγγια στον αφορά την αυτονομία εναντί των κρατών μελών. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Υπουργό, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, για να μας δώσει απαντήσεις. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις σας. Υπάρχει κάποια μερική επικάλυψη στα όσα με ρωτήσατε, οπότε και θα απαντήσω κι εγώ ε, κατά κάποιο τρόπο γενικά χωρίς να τις πιάσω μία μία τις ερωτήσεις. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω σαν μήνυμα από του Συμβουλίου είναι ότι όπως και εσείς και εμείς πιστεύουμε πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Οπότε συμφωνούμε όσον αφορά το σημείο της αφετηρίας της διαδρομής για την βελτίωση της κατάστασης. Όμως θα πρέπει κανείς να προσέξει και να μην μπερδεύει το ότι υπάρχει αναγκαιότητα βελτίωση, αλλά από την άλλη μεριά ενεδρεύει κίνδυνο κάποιες δημαγωγίες και να μην καταλήξουμε επομένω στο συμπέρασμα του ότι η κατάσταση είναι αφόρητη. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι τόσο λίγο ικανοποιητική, το πούμε έτσι, η κατάσταση, όπως ίσως έμεσα προκύπτει από κάποιους ομιλησαν. Βεβαίω Βεβαίως και να πάνε υπόψη τι είπε το ελεγκτικό συνέδριο. Βεβαίως προσπαθούμε και να συγκρατήσουμε τις, ε, την ποσότητα των λαθών που υπησέρχονται, τα οποία τώρα έρχονται στο 0,5%. Άρα να είμαστε σοβαροί και να βλέπουμε τα πράγματα με τις προβληματικές τους διαστάσεις. Και βέβαια, όσον αφορά τις ε, απάτες και όσον αφορά τη χρήση των ιδίων πόρων, εκεί είναι ακόμα πιο λίγα τα λάθη, γιατί εκεί υπάρχει, όσον αφορά την ε, απάτη, ανοχή μηδενική. Άρα να μην μπερδεύουμε τα λάθη με το δόλο. Να μην καταλήγουμε στο ότι έχει κακός η διαχείριση του προπολογισμού, γιατί δεν είναι έτσι. Και επομένω, να μην αμαυρώνουμε κάποιε πετυχημένε κατά τα άλλα πολιτικέ τη Ένωση. Θα ήταν άδικο. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποια λάθη και υπάρχει τρόπος να διορθωθούν. Αυτό συζήτησε το Συμβούλιο, αναζήτησε τις ρίζες του φαινομένου, φυσικά τίποτα δεν είναι τέλειο. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας πω τι είπε σχετικά με όλα αυτά ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνεδρίου. Τι είπε για τα λάθη. Προσοχή. Πρόεδρος του Ελληνικού Συνεδρίου, δεν το είπαμε εμείς. Είπε επομένω ο πρόεδρος ότι σε πάρα πολλά θέματα που έχει εξετάσει σχέση με τα λάθη. Τα λάθη αυτά προέρχονται από την περιπλοκότητα της νομοθεσίας των σχετικών διατάξεων. Αυτά λέει ο Πρόεδρος. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι προτεραιότητα η απλούστευση. Έχουμε δε μια σύσταση που πρέπει να την ασπαστούμε. Εγώ νομίζω θα πρέπει να το, να το πούμε αλλιώ. Μην πούμε για λιγότερους ελέγχους, για απλούστευση να πούμε, για περισσότερη ευελιξία, περισσότερο δυναμισμό στα θέματα των ελέγχων. Γιατί ξέρουμε ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τον ευέλικτο, το δυναμικό, λειτουργούν οι έλεγχοι στα κράτη-μέλη. Αυτό το κάνουμε στα κράτη μας γιατί το κάνουμε και στην Ένωση. Άρα, Προ αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Τη δε ε, εβδομάδα είχαμε το Συμβούλιο Περιφερειακής Πολιτικής και εκεί επανελήφθη αυτή η προτεραιότητα το ότι πρέπει να υπάρχει απλούστευση. θέματα που όλοι στο Συμβούλιο τα αγκάλισαν κανείς, δεν είχε ένσταση. Όσον αφορά τώρα τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας, είναι απλή η θέση μας. Είναι χρήσιμες. Θα πρέπει να αποτελούν μια πραγματική δυνατότητα για όσους θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν, αλλά αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, ε, κυρίως διοικητικά, σε κάποιες χώρες που υπάρχει ευξημένη αποκέντρωση. Και στη δική μου χώρα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Γιατί υπάρχουν πολλά και πολλαπλά επίπεδα στη διοίκηση, οπότε τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι φυσικά να επιφέρουμε βελτίωση χωρίς να πάψει να υπάρχει σεβασμός προς την διοικητική παράδοση των κρατών μελών. Το μαύρο πρόβατο βέβαια σε αυτά τα θέματα δεν είναι ούτε η Ιταλία ούτε η Ισπανία Ούτε η Ελλάδα. Είναι κάποια άλλη χώρα. Ξέρετε ποια. Τέλος. Το θέμα της μεθοδολογίας. Έχουμε πολλές ρότες. Μπορούμε να ακολουθήσουμε. Πρώτα-πρώτα πάμε για απλούστευση των διαδικασιών. Γιατί επιδέχονται βελτίωση οι μέθοδοι εργασίας μας. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ένα σωρό ε, θεσμικά όργανα, θεσμικά όργανα τα οποία δουλεύουν σκληρά και θα πρέπει επομένω να προετοιμαστούμε πριν δούμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Και έτσι να βελτιώσουμε τη διοίκηση και τη διαχείριση. όσον αφορά τον κοινωνικό προπολογισμό, Κάτι άλλο τώρα, ποια είναι η πολιτική σχέση μεταξύ του Κοινοβουλίου και των εθνικών πολιτικών αρχών. Εδώ τώρα έχουμε βέβαια και κάποια θέματα, κάποια καινούργια ζητήματα που έχουν ανακύψει, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τι σχέση θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις Εθνικές Αρχές λαμβάνοντα υπόψη και τι κοινοτικέ ε, και τις συνθήκες του Ευρωπαϊκού Ένωση αλλά και τα εθνικά συντάγματα. Εδώ τώρα βέβαια δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. και να δούμε ποιοι θα είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, τι... θα είναι οι καινούργιες ισορροπίες. βεβαίω και δεν μπορώ παρά να σα ευχαριστήσω για τα όσα είπατε. Νομίζω ότι ο διάλογος ήταν ε, πάρα πολύ και επιμένω ότι εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, τα θύματα προς τα εμπρός. θα συνεργαστούμε για την καλύτερη διαχείριση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει το ΕΚΟΦΕΝ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος μας, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση, η οικονομική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να φτάνουμε σε υπερβολές. Άλλο κριτική και άλλο αμφισβήτηση ολόκληρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οι πολιτικές αυτές λειτουργούν και λειτουργούν με τρόπο λογικό. Άρα, θέλουμε να δουλέψουμε με τρόπο επικοδομητικό, χωρίς υπερβολές και εδώ θέλω να κλείσω την παρέμβαση με αυτό το σχόλιο. Ευχαριστώ το Συμβούλιο που εκπροσωπεί του Υπουργό τον κύριο Κάνιο. Και πάμε στο σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως απαλλαγή 2008 Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τρίτο τμήμα είναι παρόν και ο Επίτροπος κ. Σαμέτ θα έρθει Επίτροπος Αν και Άντορ σε λίγο θα, σας δώσω το, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Λιμπεράτσκι σε αυτή τη φάση να μας κάνει μια παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Υπουργός μάλιστα μας παρουσίασε την όλη εικόνα. Εκαλύφθησαν πολλά από αυτά που ήθελα να πω, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πτυχές από αυτές που έθιξε ο Υπουργός. Πρώτα απ' όλα, δεν μιλάμε για κάποια απάτη, δεν αναφέρεται καμία απάτη στην έκθεσή μου όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού 2008. Ας είμαστε ξεκάθαροι στον αυτό το θέμα. Ούτε λέμε τίποτα για αμφισβήτηση ασδήποτε πολιτικής, γεωργικής πολιτικής ή πολιτικής συνοχής. Μιλάμε για τα αποτελέσματα και για το κόστος αναφερόμαστε σε δημοσιονομική πειθαρχία και το χρόνο ε, εφαρμογής υλοποίησης των διαφόρων οικονομικών μέτρων. Θα ήθελα να τονίσω ότι λέμε ότι η κατάσταση βελτιώνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη, όμως ε, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις που αναφέρονται στην έκθεση. Μία από αυτές είναι η ταχύτης. Είναι πολύ αργός ο ρυθμός. Θα χρειαζόταν 20 χρόνια και 3 μήνες με την παρούσα ταχύτητα των βελτιώσεων, τόσο ώστε ο προπολογισμό να απαλλαγεί σφαλμάτων και να φτάσουμε σε επίπεδα σφαλμάτων κάτω από 2%. Άρα ο ρυθμός είναι πάρα πολύ αργός. Και κάτι άλλο που θέλουμε να τονίσουμε, χωρίς να υπάρχει ίχνος αμφιβολίας και θα ήθελα κάποια αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας αυτό. Λοιπόν, θα να πω το ε, είναι δυνατόν μέχρι το τέλος τρέχοντος έτους να λάβουμε μια απάντηση σχετικά με την ενιαία, την ομοιόμορφη μεθοδολογία των εθνικών δηλώσεων που υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι η έκθεση υπάρχει ήδη και θέλουμε σαφείς απαντήσεις. Μπορούμε να λάβουμε σαφείς απαντήσεις. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, θέλουμε σαφή δήλωση περί της απλουστεύσεως των διαδικασιών, κυρίως στα διαθετικά ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής και θέλουμε και κάποιες απαντήσεις σχετικά με τις προκαταβολές. Τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία ήδη έχουν λάβει οι κυβερνήσεις, έχουν δαπανηθεί αυτά τα ποσά. Πώς ξοδεύτηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν για να βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση, έγινε σωστή επένδυση. Γι' αυτό έχουμε επιφυλάξει όσον αφορά το 11% το ποσοστό σφάλματος το 11% που διαπιστώνεται κάθε χρόνο. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το σφάλμα, το ποσοστό. Εξωτερικές δράσεις τώρα. Οι εξωτερικές δράσεις, εδώ το ποσοστό του σφάλματος είναι 43%, ακόμα χειρότερα. Όμως, 11% είναι το ποσοστό σφάλματος εντός κρατών μελών και εδώ νομίζω ότι μπορεί η κατάσταση να βελτιωθεί. Οι λεπτομέρειες έχουν παρουσιαστεί και θα ήθελα να μας δώσει απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πόσο χρόνο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει ένα έγγραφο. Ένα έγγραφο εργασίας το οποίο θα σκιαγραφεί σχέδια δράσης τα οποία θα είναι αξιόπιστα. Έχουμε λάβει προκαιρού κάποιο σχέδιο δράσεως. Έχει γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι δεν δόθηκε κάποια συνέχεια. Δεν έγιναν ιδέουσες βελτιώσεις. Θέλουμε το επόμενο σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα συμπεριλαμβάνει πρώτα απ' όλα σαφή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί συντονισμού εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εντός του σώματος. Θέλουμε οριζόντιο συντονισμό όσον αφορά τις δαπάνες, το, τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Δεύτερον, τι μέτρα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρονικά όρια, χρονοδιάγραμμα, κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστούν τα προτινόμενα μέτρα. Μιλώ για διαχείριση του προπολογισμού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη της. Δηλαδή, πόσο ορεύονται αυτά τα ποσά κάθε χρόνο και πώς δεν δαπανώνται όπως πρέπει. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Έχει αυξηθεί το ποσό κατά 14% το 2008 και έφτασε τα 155 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το σύστημα δεν λειτουργεί οι εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας, μεθοδολογία. Μέχρι το 2010 μπορούμε να πετύχουμε μια ενοποιημένη, μια ενιαία μεθοδολογία. Μπορεί να απαντήσετε τώρα ή χρειαζόσαστε κάποιους μήνες. Ίσως, αν αυτό ισχύει, θα πρέπει να σταματήσουμε τη διαδικασία της απαλλαγής για μερικούς μήνες μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστρέψει και δώσει απαντήσεις. Άλλο πρόβλημα που είναι πολιτικό και διοικητικό. Πολιτική και διοικητική ευθύνη της απαλλαγης για μερικους μηνες μεχρι οτι η ευρωπαικη επιτροπη επιστρεψει και δωσει απαντήσει. αλλο προβλημα που ειναι πολιτικο και διοικητικο πολιτικη και διοικητικη ευθυνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αυτο που να δούμε κάτι που αναφέρω και στην εκθεσή μου άλλωστε, είναι ότι θα πρέπει να αισθάνεται υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απομονωμένη, δεν στέκεται μόνη της. Δεν αφορά το λόγο ύπαρξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που θέτω σαν ερώτημα, είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρέπει να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει του στόχου τη. Λοιπόν, τα προγράμματα ανάκτηση. Η έκθεση δεν σας πετάει ρυθμούς, απλώς προσπαθούμε να σας δείξουμε ότι ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Ξέρουμε ποιοι ήταν οι στόχοι της χρηματοδοτήσεως, πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα, πώς τα κράτη-μέλη ωφελήθηκαν από αυτούς τους πόρους. Λοιπόν, Επίτροπε, πόσο χρόνο χρειάζεστε να σταματήσουμε τη διαδικασία της απαλλαγής, να περιμένουμε μέχρι ότου επιστρέψετε και μας δώσετε κάποια απάντηση. Διότι εμείς στο νέο κοινοβούλιο θέλουμε να ξεκινήσουμε δουλειά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να έχουμε μια σαφή βάση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θέλουμε επίσης σαφείς κανόνες όσον αφορά τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό περιμένουμε. Και οι συνάδελφοί μου πιστεύω ότι θα με υποστηρίξουν πάνω σε αυτό κυρίως οι άλλοι συγγητές. Θέλουμε ξεκάθαρη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρομαι στο σημείο 5, διότι το σημείο 5 είναι κενό. Δεν περιέχει κάτι. Να σταματήσουμε λοιπόν διαδικασία απαλλαγής. Να το κουβεντιάσουμε. Θέλουμε μια απάντηση. Ευχαριστώ. Κύριε Λιμπεράτσκι. Ο Επίτροπος Αν έχει το λόγο. Ορίστε. Mr. President, thank you. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κύριοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ευχαριστώ που μου δίνετε για πρώτη φορά στην θητεία μου την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο. Είναι ιδιαίτερη η τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα, διότι έχω και πολλά να σας υποσχεθώ. Ακούσαμε πολλά νέα για πολλά χρόνια και σωστά είπατε και εσείς και για τις αδυναμίες ε, της κοινή διαχείρισης. Αυτό με ενισχύει πολύ. Είπα τα ίδια και στην ακρόασή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είπα ότι είμαι διατεθειμένος να λάβω αυστηρά μέτρα για να καταπολεμήσω τα σφάλματα και τις καταχρήσεις επαναλαμβάνω σήμερα τη δέσμευση αυτή. Και χαίρομαι που το σχέδιο δράσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδίδει καρπούς. Το Final Impact Report για το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει και συμπεράσματα που έχουν ξεκινήσει από τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και από τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάρκεια της απαλλαγής 2006. Από τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει όλες τις δράσεις που είχε ανακοινώσει και έχει αναφερθεί και στην Επιτροπή σας και στην Ολομέλεια σχετικά με τις προόδους που επιτεύθηκαν. Άρα, εν τέλει ποια είναι τα, τα πιο σημαντικά αποτελέσματα. Τέσσερα θα σας αναφέρω. 50 έλεγχοι έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε high-risk bodies, όπου υπήρχαν δηλαδή αδύναμα ε, συστήματα διαχείρισης και επομένως μεγαλύτερη πιθανότητα σφάλματος. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να εντοπίσουμε μέρη, ε, σημεία όπου μπορεί να υπάρξουν σφάλματα. Θα συνεχίσουμε τον σημαντικό αυτό, τη σημαντική αυτή προσπάθεια ελέγχου για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον εποπτικό μας ρόλο. Δεύτερο, βελτιώσαμε τις δημοσιονομικές μας διορθώσεις. Τρίτο, ενισχύσαμε το follow-up των σφαλμάτων που εντοπίζει για το 2006 στην έκθεσή του το ελεγκτικό συνέδριο και λάβαμε τελικές θέσεις για όλες τις περιπτώσεις ανομαλιών για την διόρθωση φαρμάτων. Αυτές οι τρεις πρώτες δράσεις έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Σε τρία μόνο χρόνια βελτιώσαμε κατά 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ παλαιότερα ήταν μικρότερο το ποσό. Σε, στο σύνολο, οι δημοσιονομικές διορθώσεις από το 2000 έως το 2009 ανέρχονται σε περίπου 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις απώλειες του ε, κοινοτικού προϋπολογισμού. Τέλος, οι δημοσιονομικές διορθώσεις αποτελούν και αποτροπή για τις χώρες μέλη ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον κακοδιαχειρήσει των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι τέσσερις δράσει που αναλάβαμε και η πιο σημαντική προληπτική δράση για το 2007 2013 είναι η συμμόρφωση με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές διαχείριση με τις οποίες οφείλουν να συμμορφωθούν, όπως είπα, οι χώρες μέλη. Και αυτό πριν, από, πριν να γίνει οποιαδήποτε ενδιάμεση ε, πληρωμή. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Έχουμε τα πρώτα δείγματα ότι για το 2007-2013, για τα προγράμματα αυτά δηλαδή, ε, έχουν, οι προοπτικές έχουν βελτιωθεί. Γιατί? Διότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκαναν ελέγχους δειγματοληπτικούς επί των δηλώσεων που έγιναν μέχρι τον Μάιο του 2009. Χρησιμοποιώντας μεθοδολογία παρόμοια με του ελεγκτικού συνεδρίου, για να διαπιστωθεί το περιθώριο σφάλματος. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αποδίδουν σφάλμα που είναι σημαντικά κατώτερο από αυτό που είχε ανακοινώσει το Συμβούλιο για την περίοδο 2000-2006. Ε, Κάτι που με επιτρέπει να κοιμάμαι πιο ήσυχα. Έχουμε λοιπόν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, αν και βέβαια πρέπει να ερμηνεύονται με κάποια προσοχή. Διότι η έλεγχη, όπως είπα, ήταν δημοτοληπτική και αναφέρονταν μόνο σε 15 χώρες μέλη, διότι μέχρι τα τέλη Μαΐου 2009 δεν είχαν δηλώσει τις δαπάνες τους όλες οι χώρες μέλη. Όπως είπα, είμαστε πιο ήσυχοι τώρα. Μείωση λοιπόν του ε, περιορθωρίου σφάλματος. Συμπεραίνοντας, εγώ και ο Επίτροπος Άντορ θεωρούμε ότι τα, οι δράσεις μας αυτές έχουν αποδώσει θετικά αποτελέσματα για, και για τις τρεις προγραμματικές περιόδους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βελτιώσει τη δυνατότητά της να ε, ελέγχει και να υποπτεύει καλύτερα τη διαχείριση. Και έχουμε βάλει τα θεμέλια για να μειώσουμε το περιθώριο σφάλματος μέσω και μακροπρόθεσμα. Θεωρούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια δράσεως και οι, τα, οι πρώτοι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Ωστόσο, τονίζω ότι η δουλειά μας δεν σταματά εδώ οι δράσεις αυτές εντάσσονται πλέον στην καθημερινή μας εποπτική εργασία. Θα μου επιτρέψετε τώρα να παραδώσω το μικρόφωνο στον Επίτροπο Άντορ και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Δίνουμε το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο Άντορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα επαναλάβω αυτό το οποίο προανέφερε ο Επίτροπος Άντορ. Ότι δηλαδή για πρώτη φορά έρχομαι εδώ να σας συναντήσω. Πρώτη φορά μου δεν είναι ευκαιρία να σας γνωρίσω. Αλλά και να σας τονίσω πόσο σημαντικό θεωρούμε το να ασχολούμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως ισχύει για μένα. Γιατί μιλούμε για 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. μου ανέθεσε αυτό το χαρτοφυλάκι ο πρόεδρος Μαρόσο ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται μόνο για την απασχόληση αλλά πρόκειται και για την διαχείριση και τον σχετικό έλεγχο ενός πολύ σημαντικού ποσού γιατί τα κράτη-μέλη έχουν αρμοδιότητα διαχείριση των προγραμμάτων του Κοινωνικού Ταμείου όμως Ο τελικό υπεύθυνος για την χρηστή διαχείριση των πόρων είναι η Κομισιόν και για τους συνοτικούς μηχανισμούς. Και στη θέση που κατήχα προηγουμένως κατάλαβα, έμαθα πόσο σημαντική είναι η έλεγχη και επομένως γι' αυτό και συνεχίζω το έργο μου από αυτής της θέσεως. Όμως, χρειάζομαι την συνεργασία με του εξωτερικού οικονομικού ελεγκτέ, αλλά χρειάζομαι και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπω είπε ο κύριο Χάν, θεωρούμε ότι ο γενικό στόχο του πρόγραμματος δράση έχει μέρη επιτευχθεί. Έχουμε δε θετικά αποτελέσματα για και τις τρεις σχετικές χρήσεις. 94 έως 99 ως περίοδο προγραμματισμού έχουμε επικεντρωθεί στα των ε, διορθωτικών κινήσεων. Και αυτές οι κινήσεις αφορούν για το Ταμείο Ρωρίκη τα 864 εκατομμύρια ευρώ και για το Κοινωνικό Ταμείο και για το Ταμείο Συνοχής ε, για τις χρήσεις 8 9 1,4 δις ευρώ σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης. Όσον αφορά δε, την περίοδο 2000-2006, που σαν περίοδο προγραμματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασκήσει πιο αυστηρό έλεγχο σε συνεργασία και με τα κράτη-μέλη. Όντως ώστε να διορθωθούν τα λάθη που έχουν επισημανθεί από εμά αλλά και από το ελληνικό συνέδριο. Οπότε οι διορθώσεις φτάνουν στα 2,9 δις ευρώ για το 2008 και 9 ενώ είχαμε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την προηγούμενη οκταετία πριν δηλαδή αρχίσει να ισχύει αυτό το πρόγραμμα επίσης έχουμε ε, και την πρόθεση να διορθώσουμε τις εκθέσεις των κρατών μελών έχουμε εξυγχρονίσει, ενημερώσει τις αιτήσεις ε, εκθέσεις τόσο στην να υπάρχει προσθέμενη αξία ευρώσκα των μελών εάν υπάρχει σωστή εφαρμογή και έγκυρη εφαρμογή. Προπαρασκευαστικό έργο ήδη έχει αρχίσει όσον αφορά το κλείσιμο των προγραμμάτων 2000-2006. Έχουμε πάρα πολύ αυστηρέ διατάξει όσον αφορά την περίοδο 2007-2013 σαν περίοδο προγραμματισμού. Οπότε και ε, προχωρήσαμε σε μέτρα πρόληψη αυστηρά για συμμόρφωση των κρατών μελών, συστήματα ελέγχου, εθνικούς οικονομικούς ελέγχους, πριν έχουμε οτιδήποτε επιστροφές ενδιάμεσο χαρακτήρα, το 2006 και 2007-2013 τα πράγματα είναι, είναι απλούστερα από πολλές πλευρές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Όμως, το 2009 έχουμε περαιτέρω απλουστεύσεις για να μπορέσουμε να έχουμε για την επιλεξιμότητα διορθώσεις, μείωση των δαπανών και έχουμε επομένως για τα καταποκοπή ποσά απλούστευση για, σε σχέση με τις δηλώσεις και άλλες πληρωμές Revenue Generating Projects και εν μέρη κλείσιμο είναι θέμα το μας έχουν για να τα απλουστεύσουμε οπότε θεωρούμε ότι το πρόγραμμα δράσης έχει εφαρμοστεί. Όμως θέλουμε ο ρυθμός μας να, ο να συνεχιστεί να συνεχίσουμε την ελεκτική μας αρμοδιότητα. Να κάνουμε τις υποδείξεις για τις διορθώσεις για τη βελτίωση της αξιοποίησης των πληρώμων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος ο κ. Σεμέτα θα πάει το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις uh, του εισηγητή Λιμπεράτσκι. Καταρχάς, η παρουσία τριών επιτρόπων εδώ στη διαδικασία απαλλαγής δείχνει σαφώς ότι η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εργαστεί ως σώμα και να επομιστεί όλες τις ευθύνες σχετικά με τη διαδικασία της απαλλαγής. Και εξακολουθούμε να εργαζόμεθα τι ούτω τρόπος. Κοινή η προσπάθειά μας για να πετύχουμε τις αναγκαίες βελτιώσεις. Σχετικά με τα όσα ακούσατε σχετικά με την εκτέλεση των σχεδίων δράσης. Μας δείχνει ότι μέτρα που ήδη έχουν αναλυφθεί θα μας δώσουν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πιστεύω πραγματικά ότι δεν θα χρειαστούμε 20 χρόνια μέχρι να καταλήξουμε σε θετικό δελτίο αξιοπιστίας, σε θετική δήλωση αξιοπιστίας. Πιστεύω ότι μέσω της κοινή προσπάθειας, της προσπάθειας που θα καταβάλουμε ως σώμα, θα φτάσουμε το ταχύτερο δυνατόν εκεί. Μαζί σας. Σχετικά με το σχέδιο δράσεως. Θα θυμόσαστε ότι μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένο σχέδιο δράσεως κατά τη διάρκεια του τριμήνου που θα ακολουθήσει το διορισμό μου. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό θα συμβεί. Θα παρουσιάσω το σχέδιο δράσεως εν ευθέτω χρόνο με συγκεκριμένες δράσεις, χρονοδιαγράμματα. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Παρακαλώ, εστέ σύντομοι. Όσον θα τι ερωτήσει, πρέπει να τελειώσουμε αυτό το σημείο τη μέση διάταξη στι 5. Η κυρία Γκρέσλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Χάν. Καλώ ήρθατε. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τα καθήκοντά τη και μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε. Να σας ρωτήσω, πραγματικά παίρνετε σε σοβαρά τα μηνύματα της επιτυχίας. Εμείς βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να δούμε Πώς από τα χρήματα αυτά που ανακτώνται μπαίνουν στον προπολογισμό. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα υπόσχεται ότι θα κάνουν κάποια πράγματα τα κράτη-μέλη, ότι δεν θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα. Και όταν βλέπουμε στον προπολογισμό τι γίνεται, τα χρήματα που μπαίνουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχαν αρχικά ανακοινωθεί. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί όταν αναφέρεστε στα στοιχεία. Βλέποντας τα εθνικά ταμεία, βλέπουμε ότι με 11% επίπεδο σφαλμάτων, ατασταλίες, παραβιάσεις ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μιλάμε για 2,7 δις το χρόνο σύμφωνα το ελεκτικό συνέδριο. Και αυτό για μια περίοδο επταετή. Δεν ξέρω λοιπόν, περίπου 21 δισεκατομμύρια σύνολο. Πάνω κάτω, 20-21 δισεκατομμύρια. Αν δείτε πόσα έχουν ανακτηθεί από τα 20 δις ευρώ που κατεβλέθησαν παράνομα και τα 2,5 δις που την ίδια περίοδο επιστρέφουν, βλέπετε τι γίνεται. Μπορώ να παραθέσω και άλλα παραδείγματα. Τα κράτη-μέλη έχουν πάρει 16 δις και 1,5 δις από αυτά επεστράφησαν από τα κράτη-μέλη που πήραν τα περισσότερα χρήματα παρόλο που κάποια τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνοι για τις περισσότερες ατασταλίες. Είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί σωστά ο έλεγχος. Δεν μπορείτε να λέτε ότι λειτουργούν σωστά τα πράγματα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προσμετρήσουμε την επιτυχία βάσει των ανακτηθέντων ποσών. Ζητήσαμε να εφαρμόσει ένα νέο σύστημα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνεργασία του ελεκτικού συνεδρίου. Το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι το σύστημα δεν λειτουργεί. Τελικά πότε μπορούμε να περιμένουμε ένα σύστημα θα λειτουργεί εύρυθμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ποιο θέλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει, ποιο από του κυρίου επιτρόπου αγορεύει, βούλεται. σα ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, γνωρίζω το πρόβλημα, θα πρέπει να προσεχθεί το θέμα για αυτά τα ε, ποσά, για το θα πρέπει να είναι ορθά, ορθοί υπολογισμοί. Δεν θέλω να κάνω απρόσεκτες δηλώσεις, αλλά από ό,τι γνωρίζω, η εκτέλεση του προγράμματος δράσης οδήγησε σε βελτίωση της κατάστασης για την βιωσιμότητα αυτών των μέτρων. που βέβαια από φέτος μπορεί μόνο να σταθμιστεί. <clears throat> Είχαμε και τις σχετικές καθυστερήσεις στην περίοδο προγραμματισμού. Επομένω, ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή. Άρα και το αποτέλεσμα θα αργήσουν να έρθουν. τότε θα δούμε τα αποτελέσματα, θα δούμε τι βελτιώσεις μπορούμε να περιμένουμε όσον αφορά την ανάκτηση των πόρων. Τώρα, ο κύριος Άννα, ο Γενικός Διευθυντής, θα λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας τονίζω, πρώτα-πρώτα, ότι όταν κάποιος χρησιμοποιεί τη μέθοδο του ελληνικού συνεδρίου θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτό το οποίο μας είπαν προσέξουμε το ελληνικό συνέδριο. Ότι δεν είναι σωστό κανείς να μεταφέρει το ποσοστό λάθους σε ποσό χρημάτων. Αυτό κάνει το ελληνικό συνέδριο. Και, να κάθεται μετά τις στιγμιές ε, απόψεις της κατάστασης να τις αφρίζει. Χρονιά, τη μία χρονιά μετά την άλλη. Δεν κάνουμε μέσα εμείς. Αυτό. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να είναι το τοπίο πιο καθαρό, ούτως ώστε πρώτα πρώτα να μπορούμε ναι. να δούμε τι γίνεται μόλις κλείσει μια περίοδος με όλες τις σχετικές διορθώσεις. προσθέσαμε να δούμε μετά τις διορθώσεις τι ρυθμοί σφαλμάτων απομένουν, τι ποστολάδος τι λάθος απομενει ε, οπότε αυτό έγινε για την περίοδο 94-99. Σας είπε και ο Επιτροπός Χάν για τα αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν. Όπου τα ποσοστά ήταν κάτω από 11%. Ούτως ώστε θέλουμε αυτό να, μην, να, να έχει συνέχεια. Και πήγαμε το 2006. Μόλις γίνει το κλείσιμο βέβαια. Έχουμε επίσης ε, καλέσει τους συναδέλφους του Ελληνικού Συνεδρίου να κάτσουν μαζί μας στο ίδιο τραπέζι, να δουλέψουμε μαζί ε, για να δούμε ποια μεθοδολογία θα ακολουθήσουμε. Κάτι άλλο τώρα το οποίο έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε είναι ότι έχουμε προσπαθήσει να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σε σχέση με τις πιο πρόσφατες δαπάνες. 2007 με 2013 δηλαδή. Πέρσι προσπαθήσαμε να κάνουμε μία μήνυ δήλωση αξιοπιστία και κάνουμε ό,τι έκανε το ελληνικό συνέδριο για τα δεδομένα που τότε είχαμε. Το φθινόπωρο δηλαδή. Και έτσι να δούμε πώς είναι η κατάσταση για τις ε, δαπάνες, για τη νέα περίοδο μετά από όλες αυτές τις κινήσεις, οπότε είδαμε ότι το ποστό του σφάλματος ε, ευτυχώς είναι πολύ πιο κάτω από το 11%. Αυτό μας οδηγεί σε κάπως πιο αισιόδοξη στάση όσον αφορά το μέλλον. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Τώρα, όσον αφορά τις διορθώσεις, εδώ υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές και σενάρια. Πρώτα-πρώτα, το τι θα κάνουν τα ίδια τα κρατημέλη. Τα δε χρήματα τα οποία θα εξοικονομηθούν έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάλι ως δαπάνες από τα κρατημέλη. Γιατί θέλουμε τελικά τα χρήματα μετά τη διόρθωση να χρησιμοποιούνται για πολιτική ανάπτυξη. Άλλο σενάριο. Η Κομισιόν βρίσκει τα λάδια, το συζητάμε τα κρατημέλη, τα κρατημέλη αποδέχεται τις, τους υπολογισμούς της Κομισιόν, προβαίνει στις διορθώσεις, οπότε ούτε σε αυτήν την περίπτωση χάνονται τα χρήματα για το κράτος μέλος. Τέλος, υπάρχει περίπτωση να ανακαλύψει η Κομισιόν κάποια σφάλματα, το δέκρατος μέλος να μην συμφωνήσει με την ορθότητα των όσων λέει η Κομισιόν. Οπότε η Κομισιόν εφαρμόζει ε, την ε, τελική διόρθωση όσον αφορά τους λογαριασμούς αυτού του κράτους μέλους, οπότε χάνεται η πόρη για το κράτος και σας παραπέμπω τώρα στα στοιχεία του 2008-2009 και μιλάμε για 3,8 δις που αφορούν τις διορθώσεις που έγιναν στο όλο σύστημα κρατημέλη κομισιών από κοινό. Οπότε αυτό αντιστοιχεί και στην προηγούμενη οκταετία. Δηλαδή τότε είχαμε 3,5 δις ευρώ. Αυτά είναι τα σχέδια που έχουμε. Όποιο θέλει μπορούμε να το τα διαβιβάσουμε σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης. Αγιάλα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Και ακόμη περισσότερο ευχαριστούμε τους ε, επίτροπους που, που ήρθαν να τα συζητήσουμε σήμερα. Έχουν τρει μερούλε πριν, μόλι έφτασαν ε, αυτέ τι πληροφορίε, δεν μπορούσαμε να τι μελετήσουμε καλά για αυτό το πρόγραμμα δράση. Πάντω, θα πρέπει να δούμε για αυτό που είπε ο κύριο Υπουργό. Αν μπορούμε να έχουμε μία διαφοροποίηση, να έχουμε κάποιε περισσότερε, πιο ικανότητε πληροφορίε για το πιθανό, το ενδεχόμενο και το βέβαιο. Λάθος. Αυτό βέβαια προϋποθέτει συνεννόηση αποτελεσματική της Κομισιόν με το Ελληνικό Συνέδριο. Επίσης, αν μπορεί η Κομισιόν να μας πει δύο λόγια παραπάνω όσον αφορά την συνεργασία με το Ελληνικό Συνέδριο για να βρουν μια κοινή μεθοδολογία. Επίσης, όπως έλεγε και ο αρμόδιος για τα, τις απαλλαγής του Ινικού Συνεδρίου, το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους στη Γεωργία σε σχέση με άλλους τομείς. Τι γίνεται με τα ταμεία τι διαφορά υπάρχει στις δαπάνες. Και αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε τους νέους μηχανισμούς, ποια είναι η σχέση κόστος αποτελέσματος όσον αφορά την αύξηση των εξόδων για τους ελέγχους. Και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις για τα διορθωτικά ταμεία. Θέλει να απαντήσει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Maybe I will start and my colleagues will continue. Θα ξεκινήσω και συνεχίζουν οι συνάδελφοι. Για το τελευταίο. Κόστος ελέγχων. Σημαντικότατο. Ετοιμάζουμε ένα σύστημα που αφορά το ανοιχτό επίπεδο του σφάλματος. Θέλουμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό, το επίπεδο των δαπανών και τα ωφέλη που αποκομίζουμε. Μέσω της βαθμολόγησης θα προτείνουμε αποδεκτά ποσοστά, ανεκτά επίπεδα κινδύνου. Θα ξεκινήσει το Μάιο. Φέτος θα εξετάσουμε διάφορους τομείς πολιτικών. Σε μερικά λεπτά θα αναφερθώ στο θέμα αυτό στην παρουσίαση του προγράμματος. Ήταν το ερώτημα αφορούσε τη συνοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο και η συνοχή των μέτρων θα είναι κάτι που θα πετύχουμε το 2011 πιστεύω συνεργασία ελεγκτικού συνεδρίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργαζόμαστε στενά με το ελεγκτικό συνέδριο. Θέλω να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Αυτός είναι ο στόχος μας άλλωστε. Θετική δήλωση αξιοπιστία. Όλα τα θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεκτικό Συνέδριο, το Κοινοβούλιο, και τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργαστούν στενά. Ähm, Εγώ συμφωνώ κατά τούτο. Διεξάγονται διαρκείς συζητήσεις και με το ελεγκτικό συνέδριο για κάτι που είναι σημαντικό πρόβλημα και που διαρκώς επανέρχεται στις συζητήσεις που είναι ο όλος τομέας των δημοσίων προμηθειών. Και γι' αυτό ανέλαβα την πρωτοβουλία μαζί με τον συνάδελφό μου Μπαρνιέ να προχωρήσουμε σε στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων με στόχο μια βελτίωση στον τομέα αυτό διότι πολλά σφάλματα που διαπιστώνονται επί τόπου προέρχονται από δυσκολίες στην εφαρμογή των διατάξεων και επιθυμούμε να καταλήξουμε σε κοινέ ερμηνείε των διατάξεων αυτών από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσφέρουμε και αντίστοιχη εκπαίδευση των αρμοδίων επιτόπου. Και με τον τρόπο αυτό είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να προλάβουμε πολλά σφάλματα. Ευχαριστώ. Στάις. Τρία. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα για την έκθεση του κυρίου Λιμπεράτσκι. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή προσέγγιση. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα το έγγραφο. Περιέχει πολλά θετικά στοιχεία και θα παρουσιάσω σχετικέ τροπολογίε σε κάποια σημεία. Αν γέννη όμω, συμφωνώ μαζί σα και μπορούμε να συνεργαστούμε εξαιρετικά πιστεύω από αυτόν. Δεύτερον, να αναφερθώ στο θέμα του ελεκτικού συνεδρίου, διότι καμιά φορά κυρία ο κ. και επικρίνει το ελεκτικό συνέδριο και θα ήθελα να πω ότι και εδώ θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες, διότι πιστεύω ότι παρόλα αυτά, με την πάρο των ετών, αυτό που έκανε το ελεκτικό συνέδριο και με την εξέλιξη του ελεκτικού συνεδρίου, όσον αφορά τις αιτήσει και έκτακτες εκθέσεις, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις ακολουθούν τη σωστή ε, κατεύθυνση και συγχαίρω το ελεκτικό συνέδριο για τη δουλειά που έκανε τα τελευταία χρόνια. Η δημιουργία ενός συστήματος σηματοδοτήσεις μας δίνει μια καλύτερη εικόνα, κόκκινο φως, πράσινο φως, πορτοκαλί φως. Ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε υπάρχουν προβλήματα που υπάρχουν τα ελλείμματα των κρατών μελών, οι ελλείψεις. Έχουμε τις χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες τώρα που λαμβάνουν χώρα και δίνουν μετάλλια. Εσείς παίρνετε το χρυσό μετάλλιο, κύριε Μπονίτσι, με, για τη δουλειά που κάνατε. Θέλω να το κάνω, σαν απονείμω το βραβείο αυτό, διότι δυστυχώς τα φύγετε. Και είναι λυπηρό αυτό, διότι συνεργαστήκαμε άριστα. Τρίτον, έχουμε τρεις επιτρόπους εδώ, ανάμεσά μας. Έναν γνωρίζουμε σχετικά καλά. Μέσω της ακρόασης είχαμε και επαφές τους άλλους δύο επιτρόπους. Τους βλέπουμε για πρώτη φορά Νομίζω λοιπόν ότι ότι είναι, είναι κακά τα πνεύματα μας λένε καμιά φορά στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Σας διαβεβαιώνω ότι εμείς είμαστε καλοί, δεν είμαστε τέρατα εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Είμαστε πολύ καλοί και εργαζόμαστε σε μια ατμόσφαιρα άκρως επικοδομητική. Υπάρχουν κάποια ανώτερα στελέχη της Γενικής Διευθύνσης ΣΥΜΚΟ που μπορούν να σας το δηλώσουν αυτό. Όσον αφορά κάποιες σκληρές συζητήσεις που έγιναν κάποτε, αλλά πολύ συχνά τα αποτελέσματα των συζητήσεων είναι θετικά. Το ίδιο για την απαλλαγή. Κάνουμε την ίδια προσπάθεια. Και θέλω να θέσω στους τρεις επιτρόπους ένα ερώτημα. Διότι εκπροσωπείτε και τους άλλους 24 επιτρόπους. Θέμα. Οι δηλώσεις οι εθνικές δηλώσεις. Παράγραφος 36-42. Ο Ισπανός υπουργό ήταν ε, προηγουμένως εδώ. Αναφερθήκαμε εκτενώς στις εθνικές δηλώσεις εξοπιστίας. Πιστεύουμε στο Κοινοβούλιο ότι επ' αυτού θα πρέπει κάτι να γίνει. Θα πρέπει να στριμωχθεί το Συμβούλιο Ούτως ώστε να πάρει στα σοβαρά τις εθνικές δηλώσεις η νέα συνθήκη της Λισαβόνας το λέει στις παραγράφους 38 και 39. Η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα μέσα, ούτως ώστε να καθοδηγεί το Συμβούλιο, να το βάζει στο σωστό δρόμο. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η αντίδραση όσον αφορά τις παραγράφου 36 36-42 τις συστάσεις του κυρίου Λιμπεράτσκι που είναι σημαντικότατες θα δοθεί απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα ζητήσουμε αναβολή της διαδικασίας απαλλαγής, διότι μέσω της αναβολής της απαλλαγής μπορούμε να ασκήσουμε πίεσης και ίσως να μπουν τα πράγματα στο δρόμο τους. Αυτό είναι και το πνεύμα, νομίζω, της προσπαθίας που καταβάλει ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσει. Σε μέτα if I Πρώτα πρώτα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η απάντησή μου είναι καταφετική. Ναι, θέλω τις εθνικές ντάσεις, θεωρώ ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Να είμαστε όμως ρεαλιστές γιατί η υλοποίηση αυτής της ιδέας προϋποθέτει τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Με την συναπόφαση όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για έναν δημοσιονομικό οργανισμό που θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε την νομοθετική διαδικασία. Δεν πρόκειται μόνο για τις εθνικές ΔΑΣ, πρόκειται για πάρα πολλές και σημαντικές βελτιώσεις. Είναι κοινό μας στόχος. Αυτές οι τροπολογίες να εγκριθούν τον νωρίτερο δυνατόν. Δεύτερον, θα εξεργαστούμε μία πρόταση για την αναθεώρηση των ετησίων συνοπτικών εκθέσεων, την τυποποίηση των πληροφοριών που θα υποβάλλετε. Μελετάτε επίσης η δυνατότητα για την DAS οπότε αυτά θα είναι το βασικό μας έργο δηλαδή τη υποποίηση των όσων ζητούμε από τα κράτη-μέλη αυτόν καταλάβουν τα κράτη-μέλη με ενιαίο τρόπο να δουλεύουμε με όλους και όσον από τις γραμμές όπως έχει σήμερα το νομικό πλαίσιο υπάρχουν, τροποποιούνται, αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Είναι συστάσεις. Άρα θα πρέπει όλα αυτά εμείς να τα βάλουμε σε ένα δημοσιονομικό οργανισμό, τόσο ώστε να κρατήσει περισσότερη τάξη. Äh, ähm, Ο κ. θα συμφωνήσω με τον συνάδελφό μου και θα σας ενημερώσω ότι την προηγουμένη Παρασκευή σε ένα άτυπο Συμβούλιο Υπουργών ενθάρρυνα τις χώρες μέλη προς την, να κινηθούν προς την κατεύθυνση των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας. Γνωρίζω βέβαια το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο το οποίο επιβάλλει ορισμένα όρια. Βέβαια δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι ήδη έχουμε τέσσερις χώρες μέλη οι οποίες προβαίνουν οικειοθελώς σε αυτή την ε, δήλωση εξοπιστίας. Και νομίζω ότι είναι σωστή κατεύθυνση και για τι άλλε χώρες μέλη του Συμβουλίου. Δηλαδή τουλάχιστον να ενθαρρυνθούν να πράξουν το ίδιο. Και εκτός αυτού νομίζω έχουμε και τη δυνατότητα να καθίσουμε να σκεφτούμε και μαζί με το ελεγκτικό συνέδριο πώς ίσως είναι δυνατόν τηρουμένου του ισχύοντος πλαισίου να προβλέψουμε τέτοιες δηλώσει αξιοπιστίας και να οδηγηθούμε σε υψηλότερη αξιοπιστία. Κάτι το οποίο θα διευκολύνει το έργο μας, αλλά επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε περισσότερο με την ουσιώδη εποπτεία των ουσιωδών στόχων που θα πρέπει και αυτά να είναι βέβαια μέρη της εργασίας μας ώστε να ελέγξουμε, να εξετάσουμε κατά πόσον λειτουργούν τα διαρθρωτικά ταμεία από την πλευρά των αποτελεσμάτων και κατά πόσον δηλαδή προχωρούν προς την κατεύθυνση της Ευρώπης 2020. Κάτι που θα ήταν και μακροπρόθεσμα σωστότερη κατανομή έργου. Εντύπωση δική μου την οποία μοιράστηκα και με τους εκπροσώπους των χωρών μελών. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα τέταρτο για τέσσερις ερωτήσεις, τέσσερις απαντήσεις. Ο κύριος Οντί. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ενοχλούμε, τι να σας πω. Έχουμε προθεσμία 2 Μαρτίου, θα ψηφίσουμε 22 Μαρτίου. 2 Μαρτίου για την υποβολή τροπολογιών, έχουμε αυτές τις προθεσμίες, μερικές μέρες δηλαδή. Και σήμερα δεν ξέρω αν αυτή η Επιτροπή θα είναι σε θέση να τοποθετηθεί. Μιλάμε για θέμα αξιοπιστία στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, έναντι τη Λομελία. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή μας το κατανόησαν καλώς. Μας λένε ότι θα ετοιμάσουμε μια αντάσταση ενδιάμεση. Δήλωση εξοπιστίας. Εγώ θα το ήθελα, δεν είναι εξάρτητη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία αν υπάρχει χαμηλότερο επίπεδο που ελέγχεται από το νευτικό συνέδριο, που είναι ανεξάρτητο. Μα λένε υπάρχει σφάλμα 11%. Είναι, λένε δεν είναι 11% λιγότερο στην περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών. Δεν σα κρύπτω βουλευτή που εκπροσωπώ του πολίτε ότι δεν καταλαβαίνω πλέον τίποτα. Σα λέω αυτό που αισθάνομαι σαν ευρωβουλευτή. και πώ θα το αντιληφθούν το θέμα οι πολίτε. Είπαμε ήδη σε αυτή την Επιτροπή ότι υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας του δημοσίου χώρου. Είναι γενικό το συνέστημα ότι υπάρχει κακή διαχείριση. Βλέπουμε τι γίνεται με τα λογιστικά στην Ελλάδα κλπ. Είναι τρομακτικό. Κύριε Επίτροπε, μου λέτε ότι κοιμόσαστε καλύτερα. Ξυπνήστε όμως. Προσέξτε. να το πω και στον συνάδελφο Λιμπεράτσκι. Έκανε πολύ καλή δουλειά και λυπούμε που δεν ολοκληρώθηκε. Αλλά τον καταλαβαίνω. Διότι βλέποντα το ελεκτικό συνέδριο, τον καθηγητή Μπονίτσι, δεν ξέρω το ελεκτικό συνέδριο δίνει θετική δήλωση αξιοπιστία ή αρνητική. Εδώ και 12-13 χρόνια ήταν αρνητική δήλωση αξιοπιστία. Σήμερα τι είναι, είναι θετική δήλωση αξιοπιστία ή αρνητική. Και ω ευρωβουλευτή, ω βουλευτή, δεν γνωρίζω ποιο είναι το σωστό τεχνικό έγγραφο επί το οποίο θα μπορούμε να βασιστούμε για να ψηφίσουμε για τη θετική δήλωση εξοπιστίας. Τι περιμένουμε κύριε Επίτροπε. Μπορείτε να μας δώσετε τη διαβεβαίωση από τώρα μέχρι τις 22 Μαρτίου ότι είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε την απαλλαγή. Διαφορετικά θα αναβληθεί η απαλλαγή από ό,τι κατάλαβα. Είπε ο συνάδελφο τα πράγματα πηγαίνουν καλά, συμφωνώ κλπ. Αλλά βλέπω ότι η Επιτροπή θέλει να προτείνει μια άρνηση της απαλλαγή Ποια είναι τα στοιχεία όμως που δεν έχουμε σήμερα και που θα έχουμε στη διαθέσή μα τον Οκτώβριο. Τι αξιοπιστία θα έχουμε τον Οκτώβριο αν δεχτούμε την απαλλαγή όταν αρνηθήκαμε τον Απρίλιο, όπως κάναμε πέρσι για το Συμβούλιο, όπου την αρνηθήκαμε. Εγώ ειλικρινά ανησυχώ για τον τρόπο με τον οποίο εμείς η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού τι θα κάνουμε, κύριε Επίτροπη, κάντε σημαντική προσπάθεια από τώρα μέχρι 22 Μαρτίου. Δηλαδή, όταν θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και μετά στην Ολομέλεια, για να δώσετε διαβεβαιώσει στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού ότι μπορούμε να βασιστούμε πάνω σα, ούτε ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα. Και εξάλλου βελτιώνουν τα πράγματα. Εξάλλου θα ήταν παράδοξο, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω εδώ πέρα, ενώ τα πράγματα δεν είχαν βελτιωθεί τόσο πολύ ποτέ, όσο που έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ περισσότερο από παλιά να αρνηθεί την απαλλαγή το κοινοβούλιο. Εγώ βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Πρόεδρο, παρακαλώ, είστε σύντομοι. Ποιο θα απαντήσει. Μία απάντηση μόνο. Μία. Μην τσακωθείτε μεταξύ σα όμω, ε. Σε μέτω. Θα είμαι σύντομο. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την επίτευξη πρόοδου σε σχέση με το ότι κινήσεις για την βελτίωση της αξιοποίησης των χρημάτων της Ένωσης. Επίσης, απόψη τις προτάσεις του κ. στα κείμενά του. Εγώ, σαν ε, υπεύθυνο του χαρτοφυλακίου αυτού, θα φροντίσω να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις και συστάσεις του. Να υλοποιήσουμε τα όσα λέει και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τα κρίνετε κι εσείς από πλευρά σας. Εμείς πάντως ως Επιτροπή πρώτη θέμεθα να παρουσιάσουμε ό,τι χρειάζεται ούτως ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Dank u wel, voorzitter. Ehm, Bart Staes die had er eerder vanmiddag al over dat dit zijn elfde kwijting was. Voor mij is het de eerste. Το είπε ο κύριος Στάς Είναι η δέκατη του απαλλαγή, εμένα είναι η πρώτη. Ε, γι' αυτό ίσως είμαι τόσο αισιόδοξο. Πάντως, εγώ θεώρησα ότι και τα κρατημέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Γιατί ξέρετε, μου φάνηκε πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρο του Συμβουλίου προηγουμένως. Νομίζω ότι κρύφτηκε πίσω δηλαδή από την περιπλοκότητα των ε, διατάξεων και του καταγεγραμμένου σφάλματος. Δεν τον είδα πάντως να δείχνει πρόθεση ε, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Δεν υποσχέθηκε τίποτα. Με, φοβίζει. Και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι υπονομεύουμε την δημοσιονομική μα πολιτική. Έτσι υπονομεύουμε κάτι πολύ βασικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την αμοιβή εμπιστοσύνη. Ξέρετε, στην Ολλανδία γι' αυτό το λόγο πιστεύει ο κόσμος λιγότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα, γιατί υπάρχει δύο αντιμετώπιση όσον αφορά το κοινοτικό χρήμα. Ιδίω όσον αφορά τι λιγότερο προχωρημένε χώρε. Πάντω δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε άλλοθι αυτές τις ε, διαφορές δεν θα πρέπει να κολλάμε στα σημεία διαφωνίας θα πρέπει να δούμε πώς θα τα βρούμε, πώς θα συμφωνήσουμε και θα πρέπει να δούμε πώς θα ενεργήσουμε με υπευθυνότητα και θα πρέπει να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη επίσης να δείξουν περισσότερη προθυμία βελτίωση των πραγμάτων. Η δική μας πολιτική ομάδα θέλει να δώσει την απαλλαγή. Όμως, θεωρούμε προϋπόθεση να συνεργαστεί Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Και έτσι να μπορούμε να ασκούμε πιο υπεύθυνη πολιτική. Να προχωρήσουμε όπως είπε ο κύριος Στάς σε ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Και σας παραπέμπω και στα όσα λέει ο κ. Λιμπεράσκη στην ε, έκθεσή του όσον αφορά το εθνικό ντάς. Πώς θα γίνει να σπρώξουμε κράτη-μέλη και κομισιόν. Ορίστε, ποιος θέλει να μιλήσει. Well, I just, uh, could uh, actually... Λοιπόν, απάντησα νομίζω στο ερώτημα αυτό στα προηγούμενα σχόλιά μου. Ετοιμάζουμε την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Ετοιμάζουμε τη διατύπωση του σχεδίου κανονισμού. Σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε όσο γίνεται. όσον αφορά την πρόταση για το δημοσιονομικό κανονισμό. Μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Τι υποδοχή θα τύχει η πρόταση ο πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Δεν θέλουμε να πολεμήσουμε, δεν μιλάμε για μάχη εδώ, μιλάμε για συνεργασία να δώσουμε και κάποιο δέλεαρ πέρα των απειλών για τη βελτίωση χρήσεως των πόρων στα κράτη-μέλη. Είναι προς δικό τους όφελος, άλλωστε, να χρησιμοποιήσουν τους πόρους με τον αποδοτικότερο τρόπο. Διότι είναι χρήματα των φορολογουμένου στο κάτω-κάτω. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανησυχούν για το επίπεδο των σφαλμάτων. Υπάρχει λοιπόν η τέλεια βάση για συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Τελευταίες δύο ερωτήσεις. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ο κ. Γκάιερ έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομος. Βέβαια δεν έλαβα απάντηση. Ε, μάλλον δεν, δεν αναμένω καμιά απάντηση από τους ε, τρεις κυρίους επιτρόπους Απευθύνω χαιρετισμό άλλωστε και στους τρεις παρόντες επιτρόπους, κυρίους Σέμετα, Χάν και Άντορ. Το πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι τριπλό. Αφενός έχουμε την δήλωση αξιοπιστίας DAS, η οποία φαίνεται ασθενής. Φαίνεται ένα πράσινο χρώμα, πράσινο φως ας πούμε, για την γεωργία ε, για ορισμένε ε, χώρε μέλη. Αυτό είναι το πρώτο παράδοξο. Το δεύτερο παράδοξο γνωρίζουμε όλοι ότι τα περισσότερα χρήματα βρίσκονται σε κοινή διαχείριση και εν τέλει αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι τα ασφάλματα εντοπίζονται στις χώρες μέλη, καλούμαστε να τα διορθώσουμε και εδώ επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο κ. Γκερμπράντη. Το Συμβούλιο όμως δεν είναι απολύτως διατεθειμένο, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένο να επιμείνει ώστε να μειωθούν σημαντικά τα σφάλματα. Μας μείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει την εντολή επίσης για τον έλεγχο όπως και το Κοινοβούλιο. Και εδώ έρχομαστε στο τρίτο παράδοξο ότι έχουμε μπροστά μας τρεις επιτρόπους οι οποίοι είναι νέοι. Ε, έχουν δηλαδή και αυτοί πρόσφατα αναλάβει τα χαρτοφυλάκια τους για πρώτη φορά. Ακούσαμε ευχαρίστως τα όσα είπε ο κ. Χάν την προηγούμενη Παρασκευή και σας Πιστεύω κύριε Χάν ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Όμως ενώπιον του ερωτήματος εάν αυτό μπορώ να το θεωρήσω ως βάση για απαλλαγή ε, ε, προς την Επιτροπή αυτό μου προκαλεί ορισμένες αμφιβολίες. Μιλούμε με τρεις από εσά τώρα αλλά στην έκθεση του κύριου Λιμπεράτσκι και τον ευχαριστώ για αυτήν εντοπίζονται και άλλα σημεία σφαλμάτων που εντοπίζει ο κύριος ε, Ο υψηλός αριθμός ε, των υπαλλήλων που ε, ασχολούνται με ορισμένους τομείς και που θα θέλαμε να μειωθούν οι αριθμοί αυτοί. Με ποιον όμως θα πρέπει να συζητήσω από τους τρεις επιτρόπους. Και το γεγονός ότι έχουμε πολλά πράγματα τα οποία φαίνεται να βρίσκονται ήδη εντός του αγωγού, αλλά ακόμη δεν έχουν ε, καταλήξει. Ας δούμε εν τέλει μέχρι τον Οκτώβριο ποιες πρόοδους μπορούμε να έχουμε επιτύχει και ας δούμε μετά πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα αυτά υπό το φως αυτών των πρόοδων και τι μετά μπορούμε να προτείνουμε. Παρακαλώ, ποιος μπορεί να απαντήσει. Α, πρώτο ο κύριος Σόντεργκάρτ, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ και εγώ τους ε, τρεις νέους επιτρόπους και τους καλωσορίζω. Θα ειδωθούμε πολλές φορές τα επόμενα 4,5 περίπου χρόνια. Εγώ έχω συμμετάσχει ήδη τέσσερις φορές σε διαδικασίες απαλλαγής. Βρισκόμαστε εδώ και συζητούμε και θεωρώ ότι μπορεί να φτάσουμε ας πούμε το 2014 να συνεχίσουμε εδώ να συζητούμε, να συζητούμε για όλες αυτές τις προόδους που θα έχουν επιτευχθεί μέχρι τότε και ταυτόχρονα να έχουμε πάλι έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που να λέει ότι για τα διαθροτικά ταμεία, για τις πιστώσεις των διαθροτικών ταμείων έχουμε περιθώριο σφάλματος του τάξης του 9%. Εγώ μπορώ λοιπόν να φανταστώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και εάν αυτό συμβεί και εμείς εδώ ως ε, Επιτροπή πούμε καλά θα δώσουμε παρόλα αυτά την απαλλαγή και τότε αυτό νομίζω ότι αποδίδει το γεγονό ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που χρειαζόμαστε είναι ξεκάθαροι στόχοι. Τι θέλουμε να επιτύχουμε και με ποιο τρόπο θα επιτύχουμε του στόχου αυτού. Γιατί οι στόχοι αυτοί για μα έχουν, θα έχουν κρίσιμη σημασία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλε τι λεπτομέρειε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και την τελευταία δεκάρα πώς πανάτε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένους στόχους και να δούμε εάν αυτοί οι στόχοι πράγματι κάποια στιγμή επιτυγχάνονται. Έχω τώρα ένα ερώτημα. Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα ότι εφαρμόστηκε πλήρως το σχέδιο δράσεως. Σωστό. Νομίζω ότι θα βοηθούσε ωστόσο εάν το ελεγκτικό συνέδριο έχει την δυνατότητα να δώσει αυτό την άποψή του για τα αποτελέσματα αυτής της πλήρους εφαρμογής του σχεδίου δράσεως. Δίνω το λόγο για δύο λεπτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. έχει το λόγο. Ο Επίτροπος Χάν, να δώσω ορισμένες σύντομες απαντήσεις πρέπει κανείς να μπορεί να αντιδράσει γρήγορα, έστω και αν... Ε, ε, θα επίσης ε, για το πώς. Ο, ο συνάδελφος που ρώτησε έχει εγκαταλείψει το αίθουσα, αλλά δεν έχει σημασία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει πολύ καλή συνεργασία και με το Ελληνικό Συνέδριο. Οι υπολογισμοί μας γίνονται στην βάση της ίδιας μεθοδολογίας. Αυτό είναι ένδειξη ότι εργαζόμαστε πάνω σε μια κοινή βάση και μπορούμε να επιτύχουμε βελτιωμένα αποτελέσματα. Αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι μια ένδειξη ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και ότι αναπτύσσεται μια εμπιστοσύνη εκτός πλέον και αν αμφισβητούνται όλα τα θεσμικά όργανα αλλά νομίζω μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν που μπορέσαμε να υποβάλουμε μέχρι σήμερα νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν την βάση για να αναπτύξουμε μια εμπιστοσύνη και βασισμένη σε αυτήν την συνεργασία για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει κυρία Γκράση για τρία λεπτά το λόγο. Για Χαιρετισμούς από την Ελλάδα για εμπιστοσύνη αυτό. Σας χαιρετούμε από την Ελλάδα με εμπιστοσύνη. Αυτό είναι η απάντηση της κυρίας Γκρέσλε. Είσαστε διατεθειμένοι να βάλετε το θέμα των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας εδώ. Είσαστε διατεθειμένοι να το βάλετε αυτό το θέμα εδώ. Σας ευχαριστώ. Σκεφτείτε το και μας λέτε. Χαιρετίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Σεμέτα όσον αφορά το πρόγραμμα που αφορά τη θητεία του. Αυτή η ακρόαση ε, ε συζητήθηκε το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγινε στην Επιτροπή μου συζήτηση, γερδίζω και τον κύριο Μπονίτσι που είναι εδώ. Θα πρέπει να αναφερθεί ο κ. Σεμέντα σε πολλά σημεία, κυρίω όσον αφορά τον κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό θα αναφερθεί στο όλα, στην Όλαφ και το πρόγραμμα προτίθεται να υποβάλει στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα όσα θα κάνει στη θητεία του. Υπάρχει το πρόβλημα ε, του νέου ε, διοικητού της Όλαφ που πρέπει πολύ γρήγορα να διοριστεί. Ήδη το έχουμε συζητήσει αυτό. Θα πρέπει να εισάγεται και το θέμα του προσωρινού διευθυντή της Όλαφ. Το συζητήσαμε και πρόσφατα και καταλάξαμε πιστολές επ' αυτού και ανανέωση της Επιτροπής Εποπτείας ε, της Όλαφ. Ελπίζω να θέλετε να αναφερθείτε λίγο σε αυτά τα θέματα, σας δίνω το λόγο. Έχουμε ένα χρόνο για να τα συζητήσουμε μαζί σε αυτά τα θέματα. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Σεμέτα. Όπως σας είπα προηγουμένως, Στο μέσο επόμενο θα σα παρουσιάσω τι λεπτομέρειες ενός προγράμματος δράσης, αλλά σήμερα να σας πω ποιε είναι οι βασικέ μας προτεραιότητες για την απαλλαγή, αλλά για να συζητήσουμε αυτά τα οποία φύγετε στην επιστολή σας για την Όλαφ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη προς θεσμικές αρχές, προς τις αρχές όσον αφορά την χρηστή διαχείριση των πόρων. Αυτό και στην έκθεση του συνεδρίου αλλά και του Συμβουλίου. Και προτείνεται η χορήγηση τη απαλλαγή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά έχουν επισημανθεί κάποιοι τομείς που έχουν σχέση με τις εξωτερικές πολιτικές, εσωτερικές πολιτικές, θέματα διαχείρισης και φυσικά και με τις διαστατικές μας πολιτικές. Προτείνουμε δε, πρώτον, να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους μου, τους επιτρόπους και εγώ, ως αρμόδιος για την απαλλαγή, θα εξασφαλίσω οι συνάδελφοι να ξέρουν τι διακυβεύεται και πόσο σημαντικό είναι το να βελτιωθεί η διαχείριση των χρηματοοικονομικών συγκεκριμένα θα ενημερώνω του συναδέλφου μου για τα ζητήματα που αφορούν ε, την διαχείριση και τους οικονομικούς ελέγχους. Αυτό θα το κάνουμε όχι μόνο στις κρίσιμες φάσεις της ε, απαλλαγής, αλλά και σε σχέση με τις εκθέσει οικονομικών ελεγκτών, αλλά και των ειδικών ελέγχων. Ε, προεδρεύω μια ειδική επιτροπή, τόσο ώστε να έχουμε τη σωστή εκτέλεση ε, των συστάσεων και των ε, προτάσεων του Ελληνικού Συνεδρίου και θα βροντίσουμε να μην έχουμε ε, μη άρτια ενημέρωση και καθυστερήσεις. Θα σας ενημερώνουμε για τα βασικότερα σημεία όσον αφορά το ποσοστό του λάθους, της διορθώσεις και βελτίωση ελέγχου και γενικότερα της στρατηγικής. να αναδειχθεί η ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά τις ε, συνοπτικές εκθέσεις και να υπάρξει μέσω των δηλώσεων αξιοπιστίας ανάληψη των ευθυνών τους και να μπορέσουμε να εξηγήσουμε περισσότερο το τι θέλουμε από τα κρατημέλη για να έχουμε κάποιο είδους περισσότερη μειογένεια για τις DAS και οι αιτήσιε συνοπτικέ εκθέσει να είναι πιο αποδοτικές, να έχουν περισσότερη προσθεμένη αξία. Και αυτό να γίνει μετά από τρία χρόνια. Να υλοποιήσουμε την ιδέα της απλούστευση νομοθεσία Και στον δημοσιονομικό κανονισμό η απλούστευση αυτή και τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Συστηματική και εκτεταμένη χρήση των εφάπαξ και καταποκοπήν ποσών. Αυτό θα γίνει πέραν των μέτρων που ήδη έχουμε λάβει. Απλούστευση της διαδικασίας ανάκτησης είναι κάτι που ήδη έχει προταθεί. Θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε με κάποιο είδους ε, αιτήσει, ε, αλλά και απάντηση της αιτήσει και έγκρισή τους μέσω του ίντερνετ. μέσω μιας διαδικτυακής πύλης πιο φιλικής. Τέταρτον. Θα πρέπει να δούμε την έννοια του περιθώριου λάθος, αυτό να μπει στον δημιουργικό κανονισμό και για κάθε τομέα δαπάνης να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ελέγχου των δαπανών και ποσοστού λάθος. Μάιο 2010 επίσης θα δούμε για ενέργεια, ε, μεταφορές, ανάπτυξη της υπαίθρου, ε, μια έκθεση και κατόπιν να έχουμε εξωτερική βοήθεια, ανάπτυξη, διοικητικές δαπάνες, ε, ε, συνοχή που θα ολοκληρωθούν σαν εκθέσεις το 2011 για αυτές τις πολιτικές. Το 2012 είχαμε πει θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή. Το είχα πει όταν ήρθα εδώ για την ακρόασή μου. Τελικά όμως είπαμε με τους συναδέλφους στην Επιτροπή να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή το 2011 και το 2012. Θα εντύπουμε τις προσπαθίες μας, θα ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους να δούμε πώς θα είναι πιο αξιόπιστες, πιο ποιοτικές πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για ανάκτηση, για διορθωτικές ε, κινήσεις να έχουμε επιτόπου ελέγχους, ανάλυση δεδομένων και ε, να απευθύνουμε κάποιες συστάσεις και κάποιες ε, καμπάνιες ενημέρωσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τον πολιτή χαρακτήρα αυτών των εκθέσεων. Το συνιστά και το υλικό συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη τον πάγιο ρυθμό των λαθών. Θέλουμε επίση σε όλα αυτά να καλύψουμε και τη χρήση του 2009. Να δούμε κυρίω του τομεί που έχουν περισσότερου κινδύνου, ιδίω όσον το κλείσιμο ε, των προγραμμάτων 2000-2006 ε, στι διαστατικές δράσει και βέβαια ό,τι σφάλματα βρεθούν προ προς αυτά θα έχουμε μηδενική ανοχή και θα τα διορθώσουμε. Έκτον, θα προσπαθήσω να έχουμε πιο αποτελεσματική χρήση της αναστολή των πληρωμών δεν θα διστάσουμε να αναστήλουμε τις πληρωμές. Και όπου χρειάζεται, όταν βρούμε κενά στα συστήματα θα σταματάνε. Και ε, το δημοσιονομικός κανονισμός 2007-2011 μας το επιτρέπει αυτό. Και όλοι στην Επιτροπή θέλουμε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα όσα προβλέπετε για τους ελέγχους 2013 δηλαδή και έτσι θα εποπτεύουμε από κοντά βοηθώντας τις ε, εθνικές κυβερνήσεις εκπαίδευση των υπαλλήλων, ε, καθημερινές γραμμές, επιτόπου ελέγχους, αλλά και ανταλλαγή των αρίστων πρακτικών. Τα μέτρα που σας ανήλυσα θα βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά τα προσδεχόμενα αποτελέσματα θα έρθουν μόνο αν έχουμε ενεργή συμμετοχή όλων. Γι' αυτό προτείνω να έχουμε νέα εταιρική σχέση με τους ε, κύριους εμπλεκόμενους και κυρίως με τα κρατη Αυτή η καινούργια σχέση θα ξεκινήσει με επαφές, με συζήτηση. Κράτη-μέλη, κοινοβούλιο, ελεγκτικό συνέδριο και άλλοι εμπλεκόμενοι, όπως και οι ε, ε, αποδέκτες των πληρωμών. Να δούμε πού είναι τα προβλήματα, πού είναι τα λάθη, να συμφωνήσουμε ποια είναι η λύση. Και έτσι, με έναν αποτελεσματικό τρόπο, να διορθώσουμε τα λάθη. Να δούμε τι κάνουν οι εθνικοί ελεγκτές όσον αφορά τα, τους πόρους, κάτι το οποίο θα βοηθήσει όσον αφορά τη δήλωση εμπιστοσύνη. και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς θετικό ντάς λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και το κείμενο του κ. Λιμπάσκη για το 2008 και την απαλλαγή ούτως ώστε να έχουμε καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τις δαπάνες του κινητικού χρήματος, λαμβάνοντα υπόψη το ελληνικό συνέδριο και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την διαχείριση. να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε την πολιτική μας, να βάλουμε υπόψη το πώς κατακτήσουν τα προγράμματα, την πολιτικότητα των ελέγχων, να δούμε τον αντίκτυπο των προγραμμάτων, να δούμε πώς όλα αυτά αξιολογούνται, σταθμίζονται, αξιολογούνται και εγώ περιμένω να μας βοηθήσετε και ελπίζω ότι επί τη βάση των όσων έχουμε μέχρι σήμερα πετύχει, επί τη βάση των όσων υποσχέθηκαν η Επιτροπή, ότι το ψήφισμα για την Απαλή 2008 θα είναι ενθαρρυντικό σήμα πλευρά του Κοινοβουλίου προς την Κομισιόν. Και έτσι θα βοηθήσετε στις προσπαθειές μας να έχουμε καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση. Και έτσι να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με τους βασικούς εμπλεκομένου αλλά και τα κράτη-μέλη. Περιμένω επομένω το κείμενό σας όπου να επισημαίνετε τους τομείς που απαιτούν ε, επίγουσα δράση. Τώρα, όσον αφορά την καταπολέμηση τη απάτη, που είναι και αυτό στο χαρτοφυλακιό μου, αλλά να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον τη Όλαφ. Πρώτον, όσον αφορά τον νέο Γενικό Διευθυντή, έχουμε υποβάλει τα σχετικά έγγραφα σε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Περιμένουμε δε απάντηση. η οποία αναμένεται να φτάσει μέχρι αύριο. Και ενώ ο στόχος μας είναι το ταχύτερο δυνατόν να γίνει σχετική δημοσίευση. Και έτσι να οριστεί μόνιμα κάποιος ε, στη θέση αυτή του Γενικού Διευθυντού. Προσπαθήσαμε πως να δούμε πώς θα συνδυάσουμε τα όσα απαιτεί η κατομμύρια τη απάντηση από την Όλαφ να έχει κάποιο εμπειρία σαν εισαγγελέα σε διοικητικές αρχές να είναι κάποιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τι βαριέ ευθύνε του αξιώματο. Τώρα τον κύριο Νικάρετς που είναι ο προσωρινός γενικός στις 12 Δευτέρου του 2010 μας είπατε ότι θα πρέπει να προτείνουμε μία διαδικασία για διαβούλευση για την θέση αυτή του προσωρινού διευθυντή, διευθυντή σε σχέση και με τον κανονισμό που διέπτυλτει της ε, Όλαφ. Εγώ δεν μπορώ να σας προτείνω κάτι τώρα. Όμως, να σας πω τις ε, απόψεις μου για την κατάσταση αυτή. Η σημερινή κατάσταση, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι ο κύριος Άιλετ είναι ο προσωρινός γενικός διευθυντής. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με την αρχή της συνέχειας της διοίκησης. Από το 2005 ασκεί καθήκον πληρωτού διευθυντού, τον που είχαμε τον κύριο Μπρούνερ, και τον αντικατέστησε τότε που δυστυχώς ε, αρρώστησε βαριά. Ο κύριος Κάλλας του στείλε μια επίστοση, επιστολή συγγνώμη, και του τονίζει ότι θα πρέπει να ασκήσει τι αρμοδιότητε του με τρόπο το ώστε το Συμβούλιο αλλά και το Πρωθυπουργό Κοινοβούλιο σε τακτά διαστήματα να ενημερώνονται για τα όσα κάνει η Όλαφ. Όπω σα είπα, θα πρέπει όλα αυτά να αντικυπρωθούν ταχύτερο δυνατόν και γι' αυτό και εγώ κάνω ό,τι πρέπει. Έχουμε αυτές τις πάγιες όσον αφορά τη, την αντικατάσταση και την προσωρινή αντικατάσταση και αυτά θα ισχύσουν. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται όσον αφορά τον ορισμό επί πενταετία ενό διευθυντού. Αλλά δεν θα ισχύσει αυτή η διαδικασία για τον ενδιάμεσο προσωρινό αντικαταστάτη. Υπάρχει αυτή η νομική δυσκολία, αλλά υπάρχει και μια πρακτική ένσταση ότι δηλαδή αυτή η διαδικασία κρατάει πάρα πολύ. Οπότε αντιβαίνει στην αρχή τη συνέχεια στη διοίκηση. Αλλά είναι συνήθω πρακτική στη διοίκηση το να έχουμε ξαφνικά μια θέση κενή σε κορυφαία θέση στην ε, πυραμίδα. Άρα θα πρέπει κάποιος να αντικαταστήσει αυτόν που απεχώρησε για να υπάρξει συνέχεια. Έχουμε και ομοδεργαστή στο Συμβούλιο που ζήτησε αυτό το θέμα. Και υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση που δεν είναι έγγραφη, αλλά ε, διατυπώθηκε και από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Σας τονίζω δε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία τη Όλαφ μέσω του ορισμού του κατάλληλου διευθυντού, γιατί και το 2005 ήταν τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση, τότε που είχε λήξει η κ. Μπρούνερ. Οπότε είχε γίνει ακριβώς το ίδιο, είχε ασκήσει το κοντά του για πάνω από 9 μήνες ως προσωρινός διευθυντής και κατά αυτό το 9 μήνο αν θυμάμαι καλά είχαμε πάνω από 200 έρευνες τώρα δε σε αυτή τη φάση που έχουμε την προσωρινή ε, δίκηση ας πούμε Προσπαθούμε πάλι να λειτουργήσει με υπηρεσία βάσει της αρχής της συνέχειας. Αλλιώς, αλλιώς θα διαταραχθεί η ομαλή πορεία των ερευνών που έχουν αρχίσει και συνεχίζονται. Επίσης, Να σας πω κάτι άλλο που αναφέρει η επιστολή Κάλλας. Ο κύριος διευθυντής προτίθεται, ο κύριος Στάιλερ, να σας συναντήσει για μια ανταλλαγή απόψε. Όποτε θέλετε και τέλος, επίσης, είμαι πρόθυμος να συζητήσω οποιαδήποτε ιδέα έχετε για να βελτιώσουμε το σύστημα αντικατάστασης των διευθυντών στο μέλλον. και γενικότερα για την βελτίωση, για την αναθεώρηση του κανονισμού που διέπει τη λειτουργία της Όλαφ. Όπως ακριβώς είχε αποφασίσει και το Συμβούλιο το Φεβρουάριο 2009, είχα πει στην ακρόση μου ότι θα το θεωρήσω προτεραιότητα. Πρώτους μήνες της εντολής μου να υποβάλω ένα έγγραφο όσον αφορά τη λειτουργία της Όλαφ και την σχετική νομική βάση. Θα το υποβάλω αυτό το, αυτό το έγγραφο κάποια στιγμή πριν τις θερινές διακοπές. Περίμενα πώς και πώς επομένως να προχωρήσουμε σε διάλογο με Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Όπως προείπα. Θα ξεκινήσουμε με ένα non-paper, με αυτό το, το, το άτυπο έγγραφο που θα διατυπώνει κάποιες σκέψεις μου για να δούμε Πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε, στο Συμβούλιο, ε, εσά, να δούμε τι εναλλακτικέ έχουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να βρούμε αυτή τη συνένεση για τα πιο βασικά. Η δε πρόταση που κυκλοφορεί σε σχέση με το ψήφισμά σας, αυτά είναι η αφετηρία του προβληματισμού μας. Έχουμε διατυπώσει κάποιε προτάσει επί τη βάση αυτού του non-paper, θα κάνουμε διαβουλεύσεις με θεσμικά όργανα, να δούμε τι θα έχουμε επικοδομητικό διάλογο με εσά. Όμω έχουμε και κάποια άλλα περίπου ζητήματα όσον αφορά τη λειτουργία τη Όλαφ. Τον ανεξάρτητο χαρακτήρα τη, σχέσει με κομισιόν, σε σχέση με τον Ευρωπαίο εισαγγελέα, Όλα αυτά θα πρέπει να περάσουν από ανάλυση, να καταλήξουμε σε κάποιο μελέτη αντικτύπων και αυτά θα γίνουν στη δεύτερη φάση του προβληματισμού μας. Όσον αφορά τώρα την βελτίωση αποτελεσματικότητα τη Όλαφ, κατά την εντολή μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιώσω τι επιδόσει τη Όλαφ. Θα λάβω υπόψη τα όσα λέει η υποπτεύουσα επιτροπή, θα λάβω υπόψη το σχέδιο κειμένου του κυρίου Καζολίνο, την έκθεση της Κομισιόν, η προστασία των εγγόνων συμφερόντων της ΕΟΚ και την καβολέμηση της απάτης. Έλαβα υπόψη όλα αυτά και διαπίστωσα ότι υπάρχει ανησυχία όσον αφορά τη στρατηγία των ανθρωπίνων πόρων. Συνεργασία με τον εσωτερικό έλεγχο, την ανταλλαγή των δεδομένων, τα συνεργασία με κράτη-μέλη και όλα αυτά με την Όλαφ θα τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, όσον αφορά την νέα Εποπτική Επιτροπή, Εποπτεύουσα Επιτροπή, έχουμε καθυστερήσει όσον αφορά την ανανέωση της θητείας και θα κάνω την μπορώ του, ώστε να δοθεί όθηση και να διεκπληρωθεί αυτή η εκκρεμότητα. Και σας ενδιαφέρει το θέμα βέβαια. Επίσης, 2008-2009 έγινε μια συνεννόηση για να δούμε τι θα γίνει με τη σχετική διαδικασία. Συμφωνούμε σε κάποια θέματα, αλλά διαφωνούμε σε σχέση με το πώς και πότε θα ισχύσει η νέα διαδικασία σαν νέο εντολή των μελών τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Οπότε περιμένω πως και πως και εγώ να ανταλλάξουμε απόψει για αυτό το θέμα το νωρίτερο δυνατόν. Και σας ευχαριστώ ready to exchange views with the members of the committee. Grazie, onorevole Gressi. Ευχαριστώ κύριε Κρέσ. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την δέσμη αυτή και ευχαριστώ που είπατε και κάτι για το δύσκολο θέμα της μεταβατικής ε, αυτής Κατάληψη τη θέσεως ε, του, διευθυντού, του Γενικού Διευθυντού. Ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο σε όλη αυτή την υπόθεση. Είναι αυτέ οι ίδιε οι δικέ σα αντιφάσει. Αφενό λέτε ότι επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μα, να αναζητήσετε νέου δρόμου, Από την άλλη μεριά παραβιάζετε τα δικαιώματά μα, τα δικαιώματα συνεργασία και συναποφάσεω σε αυτή την υπόθεση του ε, ε προσωρινού Γενικού Διευθυντού από τη μια μεριά τάσεστε υπέρ των ε, δικαιωμάτων μας, από την άλλη μεριά ε, δυσχεραίνεται το έργο της ε, Όλαφ. Αυτά είναι που με ενοχλούν περισσότερο και εκεί εντοπίζω εγώ τα σημαντικότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Οι θέσεις από άποψη δικαίου είναι ξεκάθαρες και εγώ προσπάθησα να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για παιδιαρίσματα εντός εισαγωγικών, πρόκειται για την νομιμότητα της, ε, των διαδικασιών της Όλαφ. Δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά κανενός. Μου είναι αδιάφορο ποιος θα αναλάβει την διεύθυνση της Όλαφ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πόσο ανεξάρτητος θα είναι. Πόσο ανεξάρτητος θα είναι αυτός ο γενικός διευθυντής. Χρειάζεται να αναζητηθεί λοιπόν η δυνατότητα να ληφθεί μια απόφαση στο Λουξεμβούργο για ε, το θέμα αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνουν κατανοητές οι θέσεις μας. Δεν είμαι βεβαία ότι αυτό έχει επιτευχθεί. Εσείς εμένετε σε αυτήν την κατάσταση που είναι δύσκολη για όλους. Εμένετε να μην δέχεστε την χείρα που σας στείνει το Κοινοβούλιο για το θέμα της όλα. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε να ε, βρούμε ταχύε διαδικασίε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. Δεν πρόκειται να γίνει τέλειο αυτό. Θα συζητήσουμε αύριο με του συντονιστέ των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων ποια δράση θα αναλάβουμε πλέον. Εμένα θα με ενδιέφερε να μάθω τι σκέπτεται το ελεγκτικό συνέδριο του Λουξεμβούργου. Νομίζω ότι δεν είναι σκόπιμο να μην δέχεστε την χείρα βοηθείας που, που τίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που άλλωστε σας προσφέρει και την δυνατότητα να προστατευτείτε να προστατεύσετε και το Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων και εσάς προσωπικά και ολόκληρη την διαδικασία αυτή η οποία βρίσκεται, πώς να το πω, σε ανοιχτό πέλαγος αυτή τη στιγμή. Θα επαναλάβω την ερώτηση που έκανα προηγουμένως. Εάν δηλαδή είστε διατεθειμένος στην επόμενη δηλαδή δημοσιονομική αναθεώρηση και μάλιστα στο fast track το οποίο πρόκειται να έρθει γρήγορα, να ξαναθέσετε το θέμα των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε σύντομα αποτελέσματα. Αυτή νομίζω είναι και η οδός εκείνη που υπόσχεται τα περισσότερα και ταχύτερα αποτελέσματα, όπου δηλαδή μπορούμε πράγματι να βασιστούμε κάπου για να ασκήσουμε πίεση και στις άλλες χώρες μέλη. Ορίστε κύριε Επίτροπε. So I, uh, I would like to first, first of all to answer... Να απαντήσω όσον αφορά τον προσωρινό διευθυντή της Όλαφ. Συμφωνώ μαζί σας. Προς κοινών όφελος θα πρέπει αυτός ο διευθυντής, ο προσωρινός, να λειτουργεί νομικός ορθά. Και η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου έχουν τοποθετηθεί από αυτό. Έχουν την ίδια άποψη. Δεν έχει υποβληθεί γραπτός γνωμοδότηση, προφορικά τοποθετήθηκαν. Δεν του ζητήσαμε γραπτή τοποθέτηση. Πρέπει όλοι να υπομιστούμε τις ευθύνε μας. Να δούμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν διακοπεί αυτόματος ο κανονισμός για αυτόματο διορισμό σε περιπτώσεις ε, ανατέρας βίας. Χρειάζεται συνέχεια των εργασιών σε αυτό το θεσμό. Είναι βασικό στοιχείο. Και κανένας άλλος κανόνας δεν εξασφαλίζει τη συνέχιση των εργασιών, την απρόσκοπτη. Εκτός από τον αυτόματο διορισμό προσωρινού διευθυντού, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Θα το συζητήσουμε το θέμα. Στα πλαίσια του τροποποιημένου κανονισμού που πρέπει να περιέχει σαφή κανόνα σχετικό. για να αποφύγουμε παρόμοιες περιστάσεις όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. να πω εκ νέου ότι το 2005 η θητεία του κύριου Γκρούνε έληξε. και διορίστηκε σαν προσωρινός γενικός διευθυντής. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που χρησιμοποιείται και τώρα. Άρα, αν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη διαδικασία, εκείνοι που συνελήφθησαν το 2005, οι απαταιώνες, κατά τη διάρκεια του ένα μήνου, δεν θα δικαστούν και θα προσφύγουν κατά των δικών αυτών και των σχετικών διαδικασιών. Σημαντικό το ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. δεν πρέπει να αμφισβητούμε το διορισμό του προσωρινού διευθυντή. Δεν είναι κάτι που αφορά πρόσωπα εδώ αυτό που συζητούμε. Και ο συνάδελφος Μουσίμ Κάλλας που έκανε το διορισμό δεν έχουμε προσωπικά ωφέλη. Δεν είναι κάτι που αφορά το συγκεκριμένο άτομο πρέπει να καταλάβουμε το τεράστιο πεδίο δραστηριοτήτων που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Μπρούνα της ενδιάμεσης περίοδου 2005-2006 πάνω από 9 μήνο. Πάνω από 200 έρευνες παρέμειναν ανοιχτές και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Θέλουμε να αμφισβητήσουμε αυτές τις δραστηριότητε. Εγώ δεν θέλω. Ελπίζω και εσείς να μην θέλετε. Είναι προς κοινό μας όφελος να είναι η βραχυτέρα δυνατόν αυτή η προσωρινή περίοδος και να διοριστεί ο νέος μόνιμος Γενικός Διευθυντής το ταχύτερο δυνατόν. Σας παρακαλώ λοιπόν να τοποθετηθείτε σχετικά με το θέμα και το σημείο που επιβλήθη σύμφωνα με την πρότασή σας. Την πρόταση της Επιτροπής. Θα θυμόσαστε κύριε Γκρέσλε τη συζήτησή μας για το θέμα. το θέμα της, των επαγγελματικών προσόντων, του νέου Γενικού Διευθυντού κλπ. Και όλα αυτά συμπεριλήφθησαν σε ένα σχέδιο κειμένου. Στην ανακοίνωση καινής θέσεως. Και ελπίζουμε τελικά και όπως θα θυμόσαστε ξεκινήσαμε τη συζήτηση της ανακοινώσεως για καινή θέση, περί για κάλυψη θέσεως, κατά τη διάρκεια της ακροάσεώς μου, στις 12 Ιανουαρίου. Uh, Και εξακολουθούμε να ετοιμάζουμε αυτή την ε, ανακοίνωση για το για διαγωνισμό για την κάλυψη της θέσης. Πρέπει να ακούσουμε ποια είναι η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και αρχική τοποθέτηση είναι να αυξηθούν οι απαιτήσει όσον αφορά ε, τα προσόντα που θα απαιτούνται για να καλυφθεί αυτή η θέση. Και τα τρία μέρη πρέπει να συζητήσουν και οι τρεις φορείς για να εξευρεθεί κοινή λύση όσον αφορά την προκήρυξη της θέσεως αυτής. Παρακαλώ είστε γρήγοροι. Στο βαθμό του δυνατού βέβαια. Για να μπορεί να λειτουργεί σωστά η Όλαφ. εθνικές δηλώσεις, ποιο ήταν το θέμα της άλλης ερώτησης τι εθνικέ δηλώσει εξοπιστία. Λοιπόν, για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω. Για τις εθνικές δηλώσεις χρειάζεται αλλαγή του νομικού πλαισίου. Δεν απαιτεί κάτι τέτοιο το ισχύο νομικό πλαίσιο αναθεωρώντας τον δημοσιονομικό κανονισμό θέλουμε να προτείνουμε εκούσια χρήση των εθνικών δηλώσεων. Όμως και το πώς θα πρέπει να δοθούν τα κίνητρα για τα κράτη-μέλη. Κίνητρα ούτως ώστε να χρησιμοποιούν τις εθνικές δηλώσεις τα κράτη-μέλη. Όσο πιο πολύ γίνεται. Σίγουρα στο σχέδιο δημοσιονομικού κανονισμού θα προτείνουμε το θέμα αυτό της δηλώσεως αξιοπιστίας που θα ζητείτε από τα κράτη-μέλη. Και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μας υποστηρίξουν. Και αυτή η δήλωση εξοπιστίας θα επιτρέψει να είμαστε σίγουροι εμείς τα κάτι μέλη θα υπομιστούν όλες τις ευθύνες τους που απορρέουν από τον νόμο σχετικά με την χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συζητούμε γενικώ το θέμα. Τώρα θα συνεχιστεί η συζήτηση όμως. Θα συνεχίσω τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Πράγματι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία υποστηρίζουν ένθερμα τη συμπερίληψη των εθνικών δηλώσεων εξοπλισία στην εθνική του νομοθεσία, όπω είναι η Ολλανδία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία. Και θα μπορούσαμε λοιπόν να βασιστούμε σε αυτά τα κράτη-μέλη και να υποβάλουμε κάποια πρόταση για τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ντελάνσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν ήθελα να μπω στο θέμα των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας διότι πιστεύω κύριε Επίτροπε ότι είστε στο μάτι του κυκλώνα. Κάνετε κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες, θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας για να βελτιώσετε τη συνεργασία με το Συμβούλιο όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις και να εφαρμόζονται για όλους αυτά τα μέτρα. Όμως κρύβεστε πίσω από το νομικό πλαίσιο και πίσω από τη συνολική ε, ευθύνη του Συμβουλίου των Υπουργών. Και νομίζω θα έχετε προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν είστε διαθέσιμοι να είστε το πλευρό μας για αυτά τα θέματα. Ξέρω ότι πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εθνικές δηλώσεις, για να πετύχει τις εθνικές δηλώσεις. Και σαν ακροάσεις θα το είδατε αυτό. Θέλουμε να ανοίξουν οι πόρτες διάπλατα της συνεργασίας. Ήθελα όμως να μην επεκταθώ σε αυτό και θα συνεχίσω αγγλικά. Λοιπόν, για τη θέση του Γενικού Διευθυντού της Όλαφ να μιλήσω. Και σου περιπλέκω περαιτέρω τα πράγματα. Και στα σχόλια της κυρίας Γκρέσλε θέλω να αναφορώ για τις αντιφάσεις. Και βλέπω κάποιες αντιφάσεις να υπάρχουν, διότι χάρη σε πολύ βροχερό Σαββατοκύριακο στην Ολλανδία είναι 7 μέτρα το σπίτι μου κάτω από τη στάθμη θάλασσα και ανησυχούσα, όπω καταλαβαίνετε. Έβρεχε όλο το Σαββατοκύριακο. Αλλά μπορώ να κολυμβήσω. Δεν χρειάστηκε. Αλλά χάρη στη βροχή διάβαζα. Διάβαζα αυτή την προκήρυξη τη θέση και συνέκρινα όλε αυτέ τι ανακοινώσει με τι ανακοινώσει του 2004. Μια διαδικασία που παρακολούθησε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στα πίσω έδρανα. Γιατί ήμουν βοηθό τότε και βλέπω μεγάλες διαφορές μεταξύ της νέας ε, ανακοίνωσης καινής θέσεως και της παλιάς. Λοιπόν, στη νέα αυτή ανακοίνωση τι λέει. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει σημαντική επαγγελματική ε, ε, εμπειρία και εμπειρία στον τομέα το δικαστικό και στον διοκτικό τομέα. Στην παλιά ανακοίνωση πρόσκληση υποβολή ενδιαφέροντο ήταν πιο όριστη. Έλεγε ότι πρέπει να έχει σημαντική επαγγελματική ε, εμπειρία και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στον τομέα που καλύπτει αυτό το αξίωμα. Αν συγκρίνονται τα δύο, είναι το δικαστική και διοκτική εμπειρία, εισαγγελική εμπειρία, που αποκλεί εκείνο που είναι από τον τομέα επιβολή του νόμου από την αστυνομία, που είναι ένα τομέα που καλύπτει η Όλαφ. Διερωτώ με. Είπατε ότι χρειαζόμαστε σωστή ισορροπία. Το είπατε μεταξύ καταπολέμησης απάτης και ικανοτήτων διοικητικών διαχείρισης. Εδώ δεν βλέπω τίποτα όσον αφορά την εμπειρία διαχείρισης διοικητικής. Εντάξει, για καταπολέμηση την απάτη, αλλά κάποιο από, τη δικαστική, από το δικαστικό τομέα μπορεί να μην είναι ο καλύτερο διευθυντή για να χειρίζει το προσωπικό του, ο καλύτερο μάνατζερ. Και θέλουμε τον καλύτερο υποψήφιο. Όταν μιλάτε για αντιθέσει, ε, είπατε τι μα ενδιαφέρει εμά, ποιο είναι ο κοινό στόχο. Θέλουμε να είμαστε πιο γρήγοροι γίνεται στο διορισμό του διευθυντή. Ναι. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ε, ένα κοινό στόχο τουλάχιστον που θα πρέπει να είναι κοινό, δηλαδή να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό υποψήφιο. Και διαρωτώ με κατά πόσο είναι σοφό αν θέλει κανεί ένα ψάρι που είναι το μεγαλύτερο δυνατό από τη λιμνούλα, αν θα πρέπει η λιμνούλα να γίνει μικρότερη εν συγκρίση ε, με αυτά που ανακοινώναμε το 2004 για την κάλυψη θέσεω. Μήπω θα πρέπει να πάρουμε τη διατύπωση του 2004. Ξέρω ότι αποκλίνουν οι απόψεις με ενδιαφέρει εμένα αυτό το θέμα, επί μακρόν το παρακολουθούσα και σαν βοηθό και το λέω προσωπικά αυτό που λέω. Τι με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει να έχουμε καλού υποψηφίου και να έχουμε στο δυνατόν περισσότερου υποψηφίου που πληρούν κάποια κριτήρια. Και εμεί σε κοινοβούλιο τότε να δούμε ποιο τα καταφέρνει καλύτερα στην ακρόαση και ποιο δεν τα καταφέρνει να μα πείσει στην ακρόαση. Και τότε μπορούμε να καταλήξουμε στι αισθήσει μα. Ήθελα να στείλω αυτό το μήνυμα, να το διαβιβάσω προς τους, ε, στον Επίτροπο. Θέλω να ξέρω ποια είναι η άποψή του σχετικά με τη διατύπωση και κατά πόσο συμφωνεί με το στόχο ότι πρέπει να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερους καλούς υποψηφίους και να κάνουμε μια διεξοδικότατη ανάλυση αυτών και να βρούμε τον καλύτερο δυνατόν υποψήφιο. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. So, uh, uh, uh, Σε ό,τι αφορά την ε, εμπειρία ως μάνατζερ. Αυτό απαιτείται. Ε, αυτό απαιτείται στην επόμενη παράγραφο. Θα την βάλω εγώ λοιπόν μαζί, μαζί με την εμπειρία σε διώξεις κλπ. Θα ήθελα εδώ να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο για το ιδιαίτερο αυτό θέμα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε εύκαμπτοι σχετικά με τις απαιτήσει. και βέβαια νομίζω κοινός μας στόχος είναι να διοριστεί ο καλύτερος δυνατός υποψήφιος Θα ήθελα όμως να ακούσω τα σχόλιά σας, τα σχόλια της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού σχετικά με την πρόταση. Ελπίζω να λάβω και τα σχόλια του Συμβουλίου. Ήδη αυτοί έχουν υποβάλει ένα ανεπίσημο σχέδιο και νομίζω ότι θα το λάβουμε αύριο. Και μετά θα τα συζητήσουμε από κοινού και θα βρούμε ποιες είναι οι σωστές απαιτήσει για την θέση του Γενικού Διευθυντού. Ο κύριος Γκάιερ. Θα είμαι σύντομος. Θα αναφερθώ μόνο στο θέμα της Όλαφ και στις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Κύριε Σέμετα, αυτά που είπατε για τις εθνικές δηλώσεις ενισχύουν την εντύπωση που έχω ότι θα έπρεπε ίσως να περιμένει η Επιτροπή μας την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού πριν να δώσει την απαλλαγή. Για την όλα τώρα, συμφωνούμε για πολλά πράγματα. Συμφωνούμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, συμφωνούμε ότι το θέμα του διευθυντού interim προσωρινού δηλαδή θα πρέπει να είναι το δυνατόν συντομότερης διάρκειας και συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να αναλάβει το δυνατόν συντομότερο ένας γενικός διευθυντής ο οποίος να έχει προκύψει από μια απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα. Αυτό που αμφισβητείται σχετικά με την όλα τώρα είναι εάν αυτός που ε, χειρίζεται τώρα τα της Όλαφ έχει τοποθετηθεί νομίμως. Εγώ βλέπω τώρα ότι υπάρχουν δύο νομικές υπηρεσίες οι οποίες λένε ναι νομίμω, αλλά και μια νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου που λέει ότι όχι εδώ παραβιάστηκαν δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια ω βουλευτή δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή την άποψη, δεν μπορώ να πω ότι μα εδώ η ίδια η νομική μου υπηρεσία μου λέει ότι παραβιάστηκαν δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ναι, αγνώ εγώ την ε, δική τη άποψη και δέχομαι την άποψη τη νομική υπηρεσία τη Κομισιόν. Μα δεν μπορώ να τα πω αυτά τα πράγματα. Οι τρεις νομικέ υπηρεσίες, όπως άκουσα στην τελευταία ε, σύσκεψη των συντονιστών, οι τρεις νομικέ υπηρεσίες επιθυμούν να συντονιστούν στο ίδιο μήκο κύματο. Επομένω, να προκύψει μια ενιαία θέση. Με ενδιαφέρει λοιπόν εάν όντω έγινε αυτή η τριμερή σύσκεψη των ε, τριών νομικών υπηρεσιών και τι προέκυψε από αυτό. Εάν όχι, τότε θα μείνουμε εδώ όλο το βράδυ να συζητούμε ποια προσέγγιση είναι η λιγότερο επικίνδυνη. Εγώ στην σύσκεψη των συντονιστών είπα ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε την οδό που έχει τον μικρότερο κίνδυνο. Δηλαδή, εν προκειμένου να ακούσουμε την άποψη της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, η οποία βέβαια κλείνει προς την άποψη του Κοινοβουλίου, αλλά θα υπάρξουν και λιγότερες δυνατότητες, λιγότερες ευκαιρίες να υπάρξουν διαφωνίες. Σας ευχαριστώ. Έχει το λόγο. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το συζήτησε το θέμα και με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Προανέφερα και ήταν η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Είναι η ίδια με εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της νομικής υπηρεσίας. Υπήρξε, έγιναν και κάποιες συζητήσεις μεταξύ των, επι, των επικεφαλής των νομικών υπηρεσιών Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι οι θέσεις τους συγκλίνουν. Αλλά δεν συναντήθηκαν και τρεις νομικές υπηρεσίες, οπότε ίσως έτσι μπορεί να βρεθεί κοινή λύση. Δεν ξέρω αν είναι νομικός εφικτό να υπάρξει κοινή δήλωση των τριών νομικών υπηρεσιών. Ή δυνατόν, νομικός, αυτό θα ήταν ασφαλής, ασφαλέστερος τρόπος, η ασφαλέστερη λύση για τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Πρέπει να μην με παρεξηγείτε σε αυτά που λέω. Είμαι πραγματικά υπέρ των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας. Κοινό στόχο. Πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη και τη διαδικασία εγκρίσεως του δημοσιονομικού κανονισμού. αν θέλουμε να πολεμήσουμε επί σειρά ετών για το δημοσιονομικό κανονισμό, να πολεμάμε, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να βρούμε πιο ευφυή προσέγγιση όμως, ούτω ώστε να τροποποιηθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός το ταχύτερο δυνατόν. Διότι ως προανέφερα, Πολλέ τροπολογίε θα βελτιώσουν σημαντικά τον εν λόγω κανονισμό και αυτή την κατάσταση. Άρα είναι κοινόν το όφελος. Εάν περάσουν το ταχύτερο δυνατόν οι τροπολογίες. Από ό,τι ξέρω, από την κατάσταση τωρινή. Τώρα, τα περισσότερα κράτη-μέλη Ο αριθμός των 100 μελών που απαιτούνται για να περάσει δημοσιονομικό κανονισμός δεν μπορούν να συμφωνήσουν επί υποχρεωτικών εθνικών δηλώσεων. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του. Εγώ, σαν επίτροπο, θα συνεργαστώ με τα κατημέρια, αλλά και εσεί, και εσεί ω βουλευτέ, ίσω με τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να κάνετε το ίδιο. Να προωθήσετε αυτή την ιδέα μέσω εθνικών κυβερνήσεων, ούτω ώστε αυτές να, οι εθνικές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν την προσέγγιση όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστία. Κοινή δουλειά χρειάζεται. Εγώ μόνος μου δεν, θα πάρω, δεν τα καταφέρω. Και όπως σας είπα και στην ακρόαση μου, βασικός μου σκοπός είναι να πετύχω αποτελέσματα. Να έχουμε βελτιωμένο δημοσιονομικό κανονισμό που είναι προς όφελος όλων μας και όλος ιδιαίτερος προς όφελος των δικαιούχων προ οποίους οποίου απευθύνονται οι Ευρωπαϊκή Διότι αυτοί τι περιμένουν, περιμένουν σημαντικές απλουστεύσει. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Τελευταία ερώτηση, η κυρία Αγιάλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμπαθάτε με, αλλά έχω ένα κείμενο στην Επιτροπή Μεταφορών και πρέπει να φύγω σε λίγο. σε Σεμένα, μιλάμε για, το ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για βελτίωση του δημοσιονομικού κανονισμού και η αλήθεια είναι ότι όχι ως ευρωβουλευτήνα, αλλά ε, ως ειδική σύμβουλος της πολιτικής μου ομάδας είχα συμμετάσχει τότε που γεννήθηκε ο θεσμός του ΝΤΑΣ και όντας ε, ρεαλίστρια συνειδητοποίησα πόσες δυσκολίε υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη όπου είναι πιο κεντροκατευθυνόμενη η διοίκηση σε σχέση με αυτά που είναι πιο αποκεντρωμένη και ε, ακριβώς γι' αυτό οι προσπάθειές μας κατέτειναν στο να καλύψουμε ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις το να βελτιώσουν τα πράγματα που γίνεται για να υπάρξει με ρεαλιστικό τρόπο κάτι καινούργιο. Γι' αυτό και τώρα θεωρώ ότι κάτι μπορεί να γίνει, γιατί ακόμα και στη δική μου χώρα. Η δική μου κυβέρνηση κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες. Σε συνεργασία με περιφερειακές και διοικητικές αρχές, τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε διαφάνεια, να μπορούμε να αποκτήσουμε τη δυνατότητα ελέγχου και αυτοελέγχου. Και κατόπιν να σταθούν υπόλογοι μπροστά σε Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Φυσικά και θα συνεχιστεί αυτή η γραμμή πλεύσης και γι' αυτό και θα σας στηρίξουμε στις δικές σας προσπάθειες στο τι άλλο μπορεί να γίνει πέραν του ΝΤΑΣ. Τι να αυτό έχουμε ως μοναδικό Εργαλείο; για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την ητοπάθεια και την παρέτηση. Γιατί βέβαια την πρέπει να προσέξουμε γιατί είναι πάρα πολύ λεπτή χειρισμοί που απαιτείται να γίνουν σε σχέση με το DAS. Έχουμε και αυτό τον περίφημο κώδικα διοντολογίας. Ε, το, το, το είχε παλέψει ο Φουκαράς ο κύριος Μπρίνερ. Κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες. Είναι επομένω τόσο δύσκολος ο χειρισμός αυτού του, του μέσου πολιτικής που έχουμε στα χέρια μας του ΝΤΑΣ που και εγώ νιώθω κάποια απογοήτευση που δεν μπορέσαμε τότε, ο κ. Λέτκιν και άλλοι, δεν μπορέσαμε τότε να κάνουμε κάτι ακόμα πιο τέλειο. Για να έχει το Κοινοβούλιο, να έχει η Κομισιόν, η Επιτροπή μας ε, έναν τρόπο να καταλήξει στο πώς μπορούμε τελικά να εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο προσωρινός διευθυντής θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη συνέχεια στη λήψη αποφάσεων, ερευνών κλπ. έχοντας την υποστήριξη όλων. Άρα θα πρέπει να ληφθεί τελικά μια απόφαση. Αυτό να γίνει το νωρίτερο δυνατόν και γι' αυτό το λόγο να μπορέσουμε να καταλήξουμε στον καλύτερο των υποψηφίων, στον καλύτερο διευθυντή τελικά, που θα είναι μια διαδικασία επιλογής δύσκολη. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να εμπλακεί και το κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, έχετε μήπως κάποια ιδέα, έστω και προσωρινή, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια διόρθωση πορείας και το κοινοβούλιο να μπορέσει να στηρίξει συμβάλλοντας σε μια απόφαση. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στη γραμμή του πυρός. να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο υποψήφιο. Γιατί υπάρχουν εδώ κάποιες παράμετροι πάρα πολύ βασικέ, όπως η ανεξαρτησία, η αμεροληψία, η δυνατότητα προστασίας αυτών που πρέπει να προστατευτούν, αυτών που κάνουν κάποιες καταγγελίε, συγκεκριμένη πρόταση. Πολύ μακρά η ερώτηση, πολύ επιγραμματική. Ε, έληξε ο χρόνος, επιγραμματική απάντηση παρακαλώ. Ναι, θα είμαι συντομότατος. Αλλά προτείνω κάτι. Κύριος Άιλετς, ο προσωρινός διευθυντής, να έρθει. Να έρθει στο κοινοβούλιο και να μιλήσει μαζί σας. Ήδη για μερικές εβδομάδες το συζητούμε αλλά δεν μπορέσατε να τον ακούσετε τον προσωρινό διευθυντή. Νομίζω ότι έτσι έπρεπε να προχωρήσουν τα πράγματα, να προσκληθεί στην Επιτροπή και συζητήσετε μαζί του. Να δείτε πώς βλέπει αυτή την προσωρινή κατάσταση. Πώς βλέπει τις ευθύνες του. Πώς βλέπει την ανεξαρτησία του. Νομίζω ότι αυτή είναι η κανονική συμπεριφορά, η ανθρώπινη συμπεριφορά. Και συμφωνώ και με τα όσα υπόθηκαν σχετικά με την υπερβολή όσον αφορά τη σημασία των εθνικών δηλώσεων. Ναι, είναι πολύ σημαντικές. Συμφωνώ, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που θα πρέπει να επιληθούν σε αυτή την κοινή διαχείριση. Και εγώ και οι συνάδελφοί μου που είναι υπεύθυνοι για τους συγκεκριμένους τομείς, είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ας πάρουμε τις εθνικές δηλώσεις. υποτεθεί ότι είναι δεσμευτικό το μέτρο. Χρειάζεται εναρμόνιση. Χρειάζεται δουλειά. Προετοιμασία. Για να έχουμε συγκρίσιμες εθνικές δηλώσεις των κρατών μελών. Τεράστια δουλειά αυτή. Χρειάζονται προδιαγραφές ελέγχου. Οι ίδιες προδιαγραφές ελέγχου στα κράτη-μέλη προϋποθέσεις, συνθήκες. Ας μην περιοριστούμε λοιπόν σε κάποιες ιδέες, μπορεί να είναι πολύ καλές ιδέες, αλλά πιστέψτε με, υπάρχει και άλλη δουλειά πρέπει να γίνει, πολλή δουλειά, κυρίως στον τομέα της συνοχής. Ούτως ώστε να ικανοποιηθούμε όλοι όσον αφορά το ποσοστό του σφάλματος. Ευχαριστώ τον Επίτροπο κύριο Σεμέτο. Σας χαιρετίζουμε και περνάμε στο τελευταίο σημείο της Ειδική ε, έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της βοηθείας της προενταξιακής προς την Τουρκία. Δίνω το λόγο, αφού τον χαιρετήσω, στο μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Έκβιρντ, τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού γιατί μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την έκτακτη έκθεση όσον αφορά την διαχείριση της προενταξιακής ενίσχυσης αρρωγής προς την Τουρκία. Πρόκειται την πρώτη φορά που ελέγχουμε αυτή τη διαδικασία Έχουμε δύο διαφορετικά προγράμματα αρρωγή τα οποία ελέγξαμε. Πρώτον, πρώτο πρόγραμμα βοήθειας 2006 και στη συνέχεια το μέσο το προενταξιακό τη ενίσχυση που άρχισε να τρέχει αμέσω μετά. Και τα δύο προγράμματα η προενταξιακή ενίσχυση πέρασε από τη διαχείριση του συστήματος της απογεντρωμένης διαχείρισης και κατά αυτό το σύστημα δε εμείς ε, βέβαια έχουμε την γενικότερη αρμοδιότητα αλλά τα προγράμματα τα διαχειρίζονται οι τουρκικές αρχές. Οπότε και συγκρότησαν οι Τούρκοι κάποια ειδικά όργανα, κάποιες ειδικέ υπηρεσίες και τις διεπίστευσαν προς εμάς το 2003 και στα πλαίσια του συστήματος αυτού έχουμε μια αντιπροσωπεία στην ε, Κομισιόν και κάνουμε κάποιο είδου ε, εκ των προτέρων ελέγχους για διαγωνισμούς και ανάθεση συμβουλέων. Η δε ευεργετούμενη κάθε φορά είναι κάποια υπηρεσία η οποία προτείνει κάποιες ιδέες, τάσει κάποιες προϋποθέσεις και μετά διαχειρίζεται το πρόγραμμα. 500 εκατομμύρια ευρώ διατηρηθεί ετησίω για πιστώσει υποχρεώσεων. Το θέμα ήταν το κατά πόσον αυτή η πρωταξιακή αρρωγή είχε την σωστή διαχείριση από την Κομισιόν. Προσέξαμε ιδίω τρει τομεί για αυτόν τον έλεγχο πρώτα-πρώτα. Τη χάραξη αυτών των ετησίων προγραμμάτων, τη σχετική αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού Δεύτερον, το κατά ήταν το σύστημα εκτέλεσης αποτελεσματικό και τρίτον, κοιτάξαμε κάποια έργα και projects δειγματοληπτικά για να δούμε τι έγινε. Τι αδυνατά σημεία υπήρχαν στον προγραμματισμό και στη διαδικασία της εκτέλεσης. Πριν φτάσω στα συμπεράσματά μας, Πρέπει να σας πω ότι συνεργαζόμαστε και ελέγχουμε, ελέγχουμε την Κομισιόν, όχι την Τουρκία. Οπότε δεν λάβαμε υπόψη το κατά πόσο είναι έτοιμη η Τουρκία να μπει στην Ένωση. Οπότε είδαμε τι διαχείριση έγινε από πλευρά Κομισιόν. Για το πρώτο πρόγραμμα, το προενταξιακό, ελέγξαμε τι έγινε 2002 με 2006. Εντοπίσαμε προβλήματα τα οποία τα έχουμε εντοπίσει και σε άλλα προ, προγράμματα. Καθυστέρηση, κακή εφαρμογή, κακή εποπτεία και αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, είδαμε ότι δεν τέθηκαν σαφώς προτεραιότητες για το πού θα πάνε τα χρήματα. Και όσον αφορά το αποκεντρωμένο σύστημα εφαρμογή, είδαμε ότι οι τουρκικέ υπηρεσίε είχαν περάσει από έγκριση από την Κομισιόν, αλλά δεν είχαν επαρκέ προσωπικό. Σε αυτή την πρώτη περίοδο 2002-2004. Και έτσι δεν κατευθυνόταν να εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα εγκαίρως, αυτά που θα πανε τα χρηματα και οσον αφορα το αποκεντρωμενο συστημα εφαρμογη ειδαμε οτι οι τουρκικε υπηρεσιε ειχαν περασει απο εγκριση απο την κομισιον αλλα δεν ειχαν επαρκε προσωπικο σε αυτη την πρωτη περιοδο 2002 2004 και ετσι δεν κατευθυνοταν να εφαρμοστουν αυτα τα προγραμματα γερος αυτα που εμείς ελέξαμε όμως το οποίο είναι πάρα πολύ αξιοπερίεργο. Το σύστημα εξασφάλισε ότι τα προγράμματα τελικά πέτυχαν τους στόχους τους. Σε μεγάλο βαθμό θεωρούμε ότι αυτό έγινε γιατί οι τουρκικές αρχές προσπάθησαν πάρα πολύ καλά. Ε, ε, το κατόπιν είχαμε επιφέρει κάποιε αλλαγέ, αλλά βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον για να δούμε ποιε θα είναι οι επιπτώσει. Επίση, η Κομισιόν πρότεινε κάποια μέτρα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τα δύνατα σημεία όσον αφορά τα, τα, τα, τα κενά στι υπηρεσίε αυτέ, ε, τις τουρκικές, αλλά θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι έγινε όταν αυτά τα μέσα αρρωγής ε, προχωρήσουν προς εκτέλεση τα επόμενα χρόνια. Επίσης ε, καταλήξαμε στο ότι η Κομισιόν δεν είχε αρκετέ ε, πληροφορίες ώστε να προβάλλει κάποια, κάποιες ενέργειες αποτελεσματικές με αυτά τα προγράμματα. Και έτσι να πιάσουν τόπο τα κοινωνικά χρήματα. Εμείς ακριβώς για αυτό το λόγο προτείναμε κάποια, κάποιες ιδέες για να γίνει πιο αποτελεσματική η Κομισιόν. και να πιάσει τόπο το πρόγραμμα της ενίσχυσης της Τουρκίας. Βασικά, είπαμε ότι θα πρέπει να επισημανθεί πού χρειάζονται τα χρηματικά τόπινα να τα στοχοθετούμε. Ε, αντίληψη του τι, τι χρειάζεται πλευρά των αρχών και παρακολούθηση του πόσο καλά εκτέλεσε και ένα πρόγραμμα. Κάναμε ένα σωρό λοιπόν έλεγχε όσον αφορά ε, το, το, πόσο βοηθάμε, πόσο βοηθάει η Κομισιόν της υποψηφής χώρα, ε, Τα σε έλεγχοι θέλουν να βελτιώσουν ε, τα μέσα της πολιτική μας και γι' αυτό και θα πρέπει να σα τονίσω ακόμη μια φορά ότι ε, το, το, πόσο προσπάθησαν οι Τούρκοι ήταν βασικός παράγοντας ώστε να πετύχει ε, το πρόγραμμα αυτό και έτσι να βοηθηθεί η χώρα να μπορέσει να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπενχάγης. E και έτσι να μπορέσει να προσχωρήσει στο κοινωτικό κεκτημένο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάιπερ, Πίπερ μάλλον, ο συγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για αυτά που είπε. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η έκθεση είναι η βάση για την ε, απαλλαγή του 2008 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή την προενταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία 2000-2006 στα πλαίσια των μέσων που χρησιμοποιούνται και τα οποία αξιολογούνται από το ελεκτικό συνέδριο. Θα ήθελα να συνοψίσω την αξιολόγηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θεωρεί λοιπόν ότι δεν υπήρξαν σχεδόν δεν υπήρξαν προβλήματα όσον αφορά τη χρήση των πόρων. Όμως δεν καθορίστηκαν προτεραιότητες. Äh, λοιπόν, θα έπρεπε να συμμορφωθεί με τη μεταρρύθμιση του 2007 και δεν έγινε σωστέ μεταρρυθμίσεις για να γίνει ικανοποιητική αξιολόγηση προσμετρήσιμη. Ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η προσέγγιση όσον αφορά τις πιστώσεις των 200 εκατομμυρίων το χρόνο που είναι περίπου 1 δις ευρώ συνολικά, 900 ε, εκατομμύρια ευρώ στην πραγματικότητα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η προενταξιακή βοήθεια δεν καθορίστηκε σαφώς. Οι στατηγικές προκλήσεις, οι στόχοι δεν ήταν τόσο συγκεκριμένα για να προσμετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που δρομολογήθηκαν. δεν είχε τι αναγκαίες πληροφορίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει το ελεκτικό συνέδριο, για να προσμετρήσει την αποτελεσματικότητα της ενισχύση. Όλα αυτά δεν τα εφευρίσκω εγώ, αυτά είναι ε, αναφορές στο κείμενο και έχω προβλήματα να τα δεχτώ όλα αυτά και από πλευρά θετική θα ήθελα να πω ότι τα προγράμματα τα οποία αξιολογήθηκαν ήταν εντάξει. Αυτά τα προγράμματα δεν είχαν καμία ε, σχέση με την ένταξη. Ε, ήταν προγράμματα που υποστήριζαν τις τουρκικές αρχές για την καταπολέμηση της διαφθοράς το επίπεδο διαφθοράς είναι διαφορετικό από ό,τι στα Βαλκάνια, αλλά δράσαμε κάπως αυθαίρετα. Γιατί αυτά τα προγράμματα δεν συσχετίζονται με την πρόοδο προς την ένταξη, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν μπόρεσε να προσμετρήσει, να αποτιμήσει τα προγράμματα για να δει κατά πόσο υπάρχει σχέση μεταξύ των προγραμμάτων και της προσπάθειας για ένταξη. Ε, είναι αποφασιστική σημασία αυτό εγώ δεν έχω οριστική τοποθέτηση και θα ήθελα να βαθύνω στο θέμα. Έχω τρει συστάσει, λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε τι συστάσει να συμπεριλάβουμε στο ψήφισμα σχετικά με την απαλλαγή που παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, έλεγα τρει συστάσει. Πρώτα απ' όλα, οι πιστώσει του ΙΑΠΕ αφορούν προγράμματα που σχετικά με την προσχώρηση, την ένταξη, θα πρέπει να καθορίζονται περιοριστικές προτεραιότητες είναι κάτι που συστήνει το ελεκτικό συνέδριο και με το οποίο συμφωνούμε. Δεύτερον, από τη στιγμή που δεν βλέπουμε πρόοδο και δεν καταγράφονται τέτοιε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι θα δαπανούμε πολλά χρήματα και εγώ θα πρότεινα να επανέλθουμε στο ποσό του 2006, να μειωθεί λοιπόν η προενταξιακή βοήθεια. Μπορούμε να τον βιβασμό, να πούμε αυτές οι πιστώσεις προβλέπονται, και να τα βάλουμε στο αποθεματικό. Από τη στιγμή όμως που θα δούμε να σημειώνεται πραγματική πρόοδος, τότε θα απελευθερώσουμε το αποθεματικό. Αυτή είναι μια δεχόμενη λύση. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε στρατηγικά ελλείμματα και να προσπαθούμε να τα σταθμίζουμε συνεχώς. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η καλή λύση. Ε, τρίτη πρόταση, η προταξιακή βοήθεια θα πρέπει να καθοριστεί εκ νέου. Το μέσο θα πρέπει να σχεδιαστεί εκ νέου ανεξάρτητα από την περίπτωση της Τουρκίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας άμεσος αυτοματισμός μεταξύ προενταξιακής βοηθείας και της ίδιας της εντάξεως μιας χώρας. Τι γίνεται σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε άλλες μορφές, άλλους τρόπους σχέσεων γειτονίας ή συνεργασίας ενισχυμένες δεν πρέπει πάντα να καταλήγουμε στην προσχώρηση και στην ένταξη. Θα πρέπει αυτές λοιπόν οι τρεις συστάσεις να ληφθούν υπόψη, είναι σημαντικές. Να αρκεστούμε τώρα στα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήταν μια ωρεοποίηση των προγραμμάτων, των προβλημάτων, συγγνώμη, θα κάνουμε τις δέουσες, ε, πραγματοποιήσουμε τις δέουσες επαφές, θα προσπαθήσω να συνομιλήσω με τους διάφορους ενδιαφερομένους και θα προσπαθήσω στην πρώτη ψηφίσμα να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία τα οποία θα ήθελα να σας παραθέσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι τραγική για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η έκθεση διότι, για να δούμε περί τίνος πρόκειται, δεν έχουμε εδώ κάποιο είδους ε, αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Εδώ το θέμα είναι κατά πόσον μπορούμε να αποτιμήσουμε κατά πόσον έπιασαν το τα χρήματα, αν πήγαν εκεί που έπρεπε. Και αν κάτσει κανείς και διαβάσει το κείμενο του συνεδρίου, θα δει ότι υπάρχουν θέματα εδώ σημαντικά. Εκκρεμούν ερωτήματα Εωρούνται. Και εγώ έχω πολλά ερωτήματα. Θυμάμαι τον Ιανουάριο του Σουηδικού Ραδιόφωνο έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ όσον αφορά την ε, βοήθεια προς την Τουρκία. Αυτή η ενίσχυση δίνεται για να βοηθήσει την υποψήφια χώρα να ανταποκριθεί στα όσα απαιτούνται για να μπει στην ΕΟΚ. Και βεβαίω το πάρα πολύ βασικό το ότι θα γίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κριτήρια γενικά της Κοπενχάγης. Και τι πρόκειψε αυτό το ρεπορτάζ της Σουηδικής Ραδιοφωνίας. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να διαπιστωθεί το τι έγινε με τα αποτελέσματα και τι έγινε με τυχόν απάτες. Δεν υπήρχαν αποτελέσματα. Έγινε διασπάθηση του χρήματος. Επίτηδες είπαν ότι τα χρήματα αυτά πήγαν σε πολιτικές πρωτοβουλίες. Αυτά έκανε η, τότε κυβέρνηση. Το ΑΚΠ ήταν το κόμμα. Και φυσικά εκεί που είχε δύναμη κουρδική, κάποια κουρδική παράταξη, ε, το ΠΚΚ δεν δώσαν δεκάρα. Άρα, αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Δεν είναι καν θέμα το ότι δεν πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Επομένω δεν έγινε αυτό που έπρεπε, δηλαδή να βοηθήσουμε την Τουρκία να μπορέσει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να μας εξηγήσει η Κομισιόν. Επομένω, αν μπορεί να μα εξηγήσει η Κομισιόν. Τι έγινε. Τι, τι σκεφτήκαν όταν διάβασαν την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Σμιτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα επισημάνω το ίδιο με τον τον συνάδελφο. Και Θέλω να μπει στην Ένωση η Τουρκία. Όμως θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Δεν συμφωνώ με αυτό που ο κύριος Πίπερ, ότι ίσως χρειάζονται λιγότερα χρήματα, όχι περισσότερα χρειάζονται, αλλά θα πρέπει να σεβαστούν τις κοινές διατάξεις και θα πρέπει να είναι πιο αυστηροί όσον αφορά αυτά τα οποία επιτάσσουν οι κανόνες γιατί σε ορισμένε χώρες αυτά τα επιχειρήματα τα χρησιμοποιούμε τόσο ώστε να μπλοκάρουμε το δρόμο προς τη χώρα τόσο ώστε να μπορέσει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτό νοθεύει την πολιτική ατζέντα, είναι κακό την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τα άλλα πάρα πολύ άρτια είναι η, η δουλειά του του, του, του συνεδριοκύρου ε, επιβεβαιώνεται δηλαδή το ρεπορτάζ που είπατε κύριε Σόντεγκαρτ που έκανε η Σουηδική Ραδιοφωνία. Αυτό που μας λείπει είναι οι απαντήσεις στα ερωτήματα, οι απαντήσεις της Κομισιόν. Φθινόπωρο του 2009 προέκυψε το ρεπορτάζ το Σουηδικό και μίλησα, ξέρετε, με τον ρεπόρτερ που ταξίδεψε στην Τουρκία και το έψαξε. Ρώτα και τον κόσμο. Πήρατε χρήματα. Με ποιο τρόπο τα πήρατε. Πολλά προβλήματα οι μηνότητες τίποτα δεν παίρνανε. Σύριοι, γυναίκες, Κούρδοι, τίποτα. Πολλά προβλήματα απαριθμούνται στο ρεπορτάζ. και ο κύριος Φάρμ και εγώ απευθυνθήκαμε στους Τούρκους και είπαν δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αν υπάρχουν έχουν επιληθεί. Ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ όμως που θέλω Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαι πάρα πολύ αυστηρός όσον αφορά τη χρήση αυτών των πόρων. Ιδάλλως αυτό είναι αντιπαραγωγικό. γιατί τελικά θα χρησιμοποιούνται ε, ή τέλο πάντων διασπαθίζονται από αυτούς που δεν θέλουν η Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, είναι πάρα πολύ καλή αφετηρία το κείμενο του συνεδρίου. Και θα πρέπει να καταλήξει στο συμπέρασμα, δεν θα πρέπει να μπει στην Ένωση η Τουρκία. Ευχαριστώ παρακαλώ να είστε σύντομοι, διότι έχουμε ακόμα 10 λεπτά μέχρι το συνεδρίο. Ο το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ευχαριστώ πρώτα τους κυρίους και κυρίες του Ελληνικού Συνεδρίου για την εξαιρετικά χρήσιμη έκθεση. Συζητούμε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την διαχείριση της προενταξιακής βοήθειας μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Κομισιόν ελέγχθηκε και ουδή άλλος. Αυτά τα είπε σωστά ο κ. Ινβέιρα και το τονίζω και εγώ. Δεύτερο, ας εξετάσουμε την έκθεση. Δεν κατανοώ την Σουηδική, ούτε παρακολουθώ το Σουηδικό ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω λοιπόν αυτά που μου λένε οι συνάδελφοί μου ότι ακούστηκαν στο Σουηδικό ραδιόφωνο και ούτε νομίζω ότι εξυπηρετεί την συζήτηση. Για δύο πράγματα, δύο πράγματα μάλλον με παραξένεψαν στην έκθεση και με ανησυχούν. Αφενός τονίζει το ελεγκτικό συνέδριο ότι για τα πρώτα χρόνια της προσέγγισης δεν υπήρχαν κριτήρια για την μέτρηση της επιτυχίας των όσων έργων προωθούνταν στην Τουρκία. Δηλαδή αυτά που συζητούσαμε σήμερα το απόγευμα για την πολιτική συνοχής προφανώς δεν τα εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια παρόμοια περίπτωση. Δεύτερο, η βοήθεια προσέγγισης, μα δεν είναι και η πρώτη φορά που την ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί λοιπόν διαπιστεύονται όργανα τα οποία είναι προφανές ότι με το προσωπικό που διαθέτουν δεν μπορούν να αποδώσουν αυτά που αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, θα πρέπει να παίξει το ρόλο του καθοδηγητού να δείξει δηλαδή ποιο είναι ο σωστό τρόπο διαχειρίσεω των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λοιπόν διαρωτώ με γιατί τα πράγματα έγιναν έτσι. Διαβάζω επίση την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της Ανατολικής Ανατολίας δεν μπορούσε να κάνει τίποτε περισσότερο διότι υπήρχε εκεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μα γιατί προσπαθεί να προωθήσει θέματα, έργα εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου δεν μπορεί ούτε τις ανάγκες να αξιολογήσει ούτε και την πρόοδο των έργων. το ότι δεν ανταποκρίνονται τα κριτήρια στα μέσα, κύριε Πίπερ, είναι, πρόβλημα της Κομισιόν. Για θέματα στρατηγικής, λοιπόν, πάλι πρέπει να μεμφθούμε την Κομισιόν και να επιμείνουμε ώστε αυτά τα πράγματα να αλλάξουν και να συνδεθούν με τα κριτήρια της σύνδεσης. Συμφωνώ, αλλά δεν συμφωνώ στο τρίτο θέμα σας. Συζητούμε εδώ έκθεση, όπως είπα πριν, του ελεγχτικού συνεδρίου για την βοήθεια προσέγγισης που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια χώρα η οποία χώρα είναι υποψήφια για ένταξη και αυτό είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει αυτό. Το ότι τα κονδύλια ΙΠΑ μπορούν να διατεθούν και για άσκηση πολιτικής γειτονίας δεν συζητείται εδώ, δεν είναι θέμα που είναι υποσυζήτηση εδώ. Ο κύριο Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα τώρα. Για μένα πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα που δείχνει ακριβώς τα όσα είπα προηγουμένως. Η πολιτική και διοικητική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτές δεν ανταποκρίνεται. Προφανώς δεν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι υπεύθυνη για τόσο σημαντικά θέματα όπως είναι αυτά της ε, προσέγγισης της Τουρκίας. Δεν φαίνεται να αισθάνεται ότι είναι υπεύθυνη για την ε, ορθή διαχείριση χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να λοιπόν ένα ακόμη σχόλιο για την απαλλαγή. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα. Ε, Εγώ, πρόεδρε, Θέλω να επαναλάβω ότι δεν κρίνεται εδώ η υποψηφιότητα της Τουρκίας. Φυσικά και αυτό έχει σημασία, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να πιάνουν τόπο τα χρήματα όσο γίνεται περισσότερο. Παρ' αυτά. Κύριε Πίπερ, μακάρι αυτά που λέει το συνέδριο όσον αφορά τα προγράμματα. Μακάρι. να είχε εφαρμοστεί γενικότερα στην πολιτική της συνοχής. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν, εδώ δεν έχουμε του δείκτε και κριτήρια που χρειάζονται τόσο ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τον το αν ήταν αποτελεσματική η αρρωγή. Και ό,τι δείκτε υπήρχαν δεν χρησιμοποιήθηκαν αρκετά από την Κομισιόν. Oh, είπαμε για των τελωνίων και Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες μεταβλητές και το επισημαίνει ότι εκεί έγινε μέτρηση αποτελεσματικότητας από το συνέδριο. Άρα το συμπέρασμα θα πρέπει να κάτσει και να θεωρήσει μια σειρά πραγμάτων η Κομισιόν. Και έτσι να συνεχίσουμε να βοηθούμε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Φιλόρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ και εγώ στην έκθεση και μόνο του ελεκτικού συνεδρίου και τα έγγραφα εργασία του κυρίου Πίπερ. Τα άλλα θέματα δεν είναι για συζήτηση σημερινή. Τρία πράγματα έχω να πω. υπήρξαν αδυναμίες, αυτό είναι σίγουρο, όσον αφορά την πρωτεξιακή βοήθεια που δόθηκε στην Τουρκία, που το 2000 ξεκινούσε από το 0. Ξέρω ότι έχουμε εμπειρία πρωτεξιακή βοηθείας για άλλες χώρες, αλλά με την Τουρκία ξεκινούσαμε εκ του μηδενός. Ήταν μια μέθοδο, περίοδος μαθητείας και για τις τουρκικές αρχές και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε πάρει μαθήματα ηρίστον παρόδο ότι διαρωτώμε ακούγοντας κάποιες παρεμβάσεις κατά πόσο αν δια... έχουμε διαβάσει την ίδια έκθεση. Στα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου δεν βλέπω ότι δεν υπήρχε καμία προτεραιότης ή καμία σχέση με τα ενταξιακά κριτήρια. Εκείνοι πήραν το λόγο, μας είπαν ότι δεν υπήρχε κάποια σχέση με τα ενταξιακά κριτήρια. Ας μου το αποδείξουν ότι υπήρχαν προγράμματα που δεν είχαν τη σχέση με τα πενταξιακά κριτήρια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Όλα τα κριτήρια, όλα τα κριτήρια, τα ενταξιακά χρησιμοποιήθηκαν ως αναφορά για όλα τα προγράμματα. Και η πενταξιακή βοήθεια για την Τουρκία πάντα το συναρτήσει κριτηρίων ενταξιακών, συναρτήσει προτεραιοτήτων εταιρική σχέσεως ενταξιακής και συναρτήσει του των MIPD που ήταν έγγραφα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για τη διοχέτευση των παρεμβάσεών μα. Ίσως να μην υπήρξε επαρκής προτεραιότητα ή προτεραιότητα να μην ήταν καλώ καθορισμένη, επαρκώ. Αλλά αυτό είναι άλλο. Πείτε μου ένα πρόγραμμα όμως που δεν συσχετιζόταν με προτεραιότητα της εταιρική σχέσεως ε, για την ένταξη τα ενταξιακά κριτήρια. Άλλη παρατήρηση. Από το 2007 εισαγάγαμε βελτιώσεις σημαντικές που αναγνωρίστηκαν εξάλλου στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Εισαγάγαμε δίκτες και κριτήρια επιλογής. Τους περίφημους δίκτες SMART και RACER που επέτρεπαν αυτοί οι δείκτες ακριβώς αυτό την καλύτερη προσμέτρηση τη σκοπιμότητα των προγραμμάτων που μα υποβαλόταν. Κανένα πρόγραμμα, κυρίε και κύριοι, δεν γινόταν αποδεκτό που δεν πληρούσε αυτά τα κριτήρια. Κανένα, λέγω. Τρίτο σχόλιο. Συμφωνούμε επίση με το ελεκτικό συνέδριο. Πράγματι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Και τώρα ετοιμάζουμε νέα προσέγγιση που θα διέπει τα προγράμματα ΥΠΑΡ. Όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά για όλες τις υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες. Στατηγική τομεακή προσέγγιση θέλουμε να αναπτύξουμε για την τομεακή υποστήριξη ξεκινώντας από την τομεακή στατηγική που παρουσιάζουν τα υποψήφια κράτη ή ξεκινώντας από τομείς που θέλουμε να υποστηρίξουμε στα υποψήφια κράτη για να δώσουμε στατηγική αξία στις προτεραιότητες και αντολισμούς της προενταξιακή μας βοήθειας. Εγώ είμαι έτοιμος να απαντήσω σε άλλε ερωτήσεις όσον αφορά το σουηδικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Εάν είχατε τυχαία συναντήσει δημοσιογράφου, δεν ξέρω, μας ερχόταν να μας δουν και χαιρόνταν που τους δείχναμε στοιχεία που τους επιτρέπουν να διεξαγάγουν έρευνα σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δύο λεπτά αν θέλετε να ολοκληρώσετε. Στον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου δίνουμε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάω το ρολόι. Τρία σχόλια. Πρώτον, σωστά υπόθηκε ότι υπάρχει επιμερισμός εργασιών μεταξύ ελεκτικού συνεδρίου και πολιτικών. Το ελεκτικό συνέδριο κοιτάει τα στοιχεία και την αποτελεσματικότητα, την οικονομία, την αποδοτικότητα των πολιτικών. Υπήρξαν επιτυχίες οι πολιτικές. Οι πολιτικοί συναγάγουν τις πολιτικές συνέπειες. Καταλήγουν συμπεράσματά τους μάλλον οι πολιτικοί. Θα πρέπει να γίνει ένα κράτος, κράτος μέλος ή όχι. Έχοντας αυτά υπόψη, έρχομαι στο δεύτερο σχόλιο μου. Σχόλιο μου. Η πρόταση του κυρίου Πίπερ από μια πρακτική σκοπιά πρέπει να πω ότι αντικατοπτρίζει πιστά την ειδική μας έκθεση. Προσθέτει όμως και τα δικά του συμπεράσματα στις προτάσεις για τα που κάνει για που κάνει δεν έχω πρόβλημα την πρόταση 1, 2, 5, 6 και 7 ή 4 είναι πολιτικής φύσεως η πρόταση. Όχι περισσότερα χρήματα στην Τουρκία. Μη τους δώσετε καθεστώς πλήρους μέλους, αλλά προνομιούχα εταιρική σχέση. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Θα πω από τοποθέτηση. Είναι θέμα πολιτικό. Τρίτον στοιχείο. Αν αντικατοπτρίζεται εδώ η ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου είναι πολύ αρνητικά. Εκφράζονται, τονίζονται τα αρνητικά στοιχεία της εκθέσεως περισσότερο και δεν είναι ισορροπημένη η παρουσίαση δεν προβάλλονται αρκετά τα θετικά στοιχεία. ο κ. της Επιτροπής το είπε αυτό. Να κλείσω λέγοντας ότι βεβαίως δεν γνωρίζω το ελεκτικό συνέδριο δεν κρίνει την πολιτική πλευρά της αποδοχής της Τουρκίας θέματα όπως κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. κλπ. Αλλά έχουμε την εντύπωση ότι η ποιότητα η διοικητική στα διάφορα τουρκικά υπουργεία είναι καλύτερη διοίκηση από ό,τι σε, σε πολλές άλλες υποψήφιες χώρες των Βαλκανίων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.